Good morning to you all. Καλημέρα σας όλοι συνάδελφοι και πολίτες. Αρχίζει η συνεδρίαση. Λοιπόν, ανακοίνωση για τις εργασίες των συντονιστών. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν ομόφωνα τις κατεπίγουσες, δύο διαδικασίες κατεπίγουσες για τις αναφορές 1357-13 και 1666 επίσης 13 θα προχωρήσουμε με κατεπήγοντα τρόπο στην εξέταση των δύο αυτών αναφορών στην ε, ημερήσια διάταξη της 16ης ε, ε, Δεκεμβρίου θα επικυρώσουμε την γραπτή διαδικασία ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει ξεκινήσει και σχετικά τώρα με την ημερήσια διάταξη της συνάντησής μας τον Ιανουάριο θα διανεμηθεί και θα εγκριθεί, θα επικυρωθεί με τη γραπτή διαδικασία όπως προβλέπετε. Μετά από αιτήματα των συναδέλφων Γιάρ και Μποστινάρου, έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα για δύο αναφορές, την 13-17 του 13 και την 40-48 επίσης του 13. Ταυτόχρονα έχουν γίνει ανακοινώσεις από πλευράς μου όπως προβλέπονται στα διάφορα της ημερησίας διάταξης. Όποιος ενδιαφέρεται, όποιο μέλος ενδιαφέρεται μπορεί να τα αναζητήσει. Επιβεβαιώθηκε επίσης η απόφαση που είχε ήδη ληφθεί για την έγκριση της συνεδριάσεως του προγράμματος της συνεδριάσεως της 16ης ε, Δεκεμβρίου έγινε δεκτή με πλειοψηφία από, την, ε, από τους συντονιστές. Δεν έχω κάτι εδώ να προσθέσω. Δίνω το λόγο στην κυρία Σντάνοκα. Θέλω να αναφερθώ στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Chiudiamo allora Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα. Και το επόμενο θέμα είναι η μερίσια διάταξη της σημερινής μας συνεδριάσεως. Προβλέπει η εξέταση της ημερησίας διατάξεως σαν βασικό θέμα την εξέταση της εκθέσεως της αποστολής στην Γαλλικία, την εξέταση των αναφορών ε, τις σχετικές με τα εξωτερικά σύνορα και τους κτηνιατρικούς ελέγχους ε, στα σύνορα. Υπάρχουν επίσης κάποιες αναφορές ε, που ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας στη Βαλένσια, πάντα της Ισπανίας. Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες αναφορές που άπτονται της συμβατότητας της ε, νομοθεσίας ε, για τις οικοδομές ε, στην Κύπρο με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υπάρχει επίσης μία αναφορά σχετικά με την πιθανή παραβίαση του κοινοτικού κανονισμού στον ανταγωνισμό στην Ελλάδα θα υπάρξει επίσης και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς μας φέτος, συνάδελφος Βαλένσα, και υπάρχουν και κάποιες επιπλέον αναφορές γύρω από θέματα διακρίσεων εις βάρος ιδιοκτητών εδαφών στην Γαλλία. Έχει προταθεί επίσης και μια αλλαγή κάποιων θεμάτων που είναι στην ημερήσια διάταξη ε, με τη σειρά την οποία θα σας παρουσιάσω. Να ξεκινήσουμε ε, με το 3, 4 και 5, κλείνοντας τα θέματα αυτά, μετά να περάσουμε στο 11 και μετά το 6, 10, 7, 8, 9, 12 προβλέπεται η παρουσία των αναφερόντων, αναφερομένων καλύτερα, για τις 11, 7, 8 και 9. Λοιπόν, δεν έχω κάποιες άλλες ε, ε, ανακοινώσεις εδώ και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Στάνοκα. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτείνω το 6 δηλαδή την εξέταση των τροπολογιών για την ε, αποστολή στη Γαλλικία. Translations of Να την αποσύρουμε. Γιατί δεν έχουμε ε, τα φράσεις των τροπολογιών. Ε, πώς να εξετάσω τροπολογίες που δεν τις καταλαβαίνω. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνω ισπανικά. και δεν τις έχω στις γλώσσες που καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, για το περιγραφικό μέρος, είχε κατατεθεί ως το τελικό έγγραφο εργασίας και υποβλήθηκε το Νοέμβριο πριν, πριν να λάβουμε την επιστολή της ΑΦΚΟ του κύριου Κασίνη δηλαδή, που μας εξηγούσε τη διαδικασία έγκρισης των αποτελεσμάτων της διερευνητικής επίσκεψης. Αυτό λοιπόν τώρα αντιφάσκει με τις συστάσεις εκείνες. Και η Αγγέλικα Βέρτμαν και εγώ Είμαστε δύο μέλη της, αποστολής, της τριμελούς αποστολής και θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε το περιγραφικό μέρος που θα έχει την άποψη της πλειοψηφίας και την πλειοψηφία ενός με δύο έγγραφα της Αγγέλικα Βέρταν και της Τατιάνας δάνο από και χωριστά από τον Φιλίπ Μπουλάν. όπως συνέστησε η ΑΦΚΟ δηλαδή, αυτό το περιγραφικό μέρος θα το υποβάλουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Διότι δεν μπορέσαμε να το πράξουμε προηγουμένως. Διότι η μόνη συνεδρίαση που είχαμε για αυτό το περιγραφικό μέρος έγινε χθες και δεν συμφωνήσαμε. Άρα πρέπει να κάνουμε γνωμοδότηση πλειοψηφία, γνωμοδότηση μειοψηφία για να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Προτείνω λοιπόν αναβολή του 6 από τη σημερινή διάταξη για την επόμενη μας συνεδρίαση. Νομίζω ότι πάνω στο συγκεκριμένο σημείο η Επιτροπή μας και οι συντονιστές έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε ψηφίσει επανειλημμένα. Δεν πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου μια συζήτηση, αλλά υπάρχει η συγκεκριμένη πρόταση της κυρίας Ντάνοκα και θα ήθελα τις απόψεις των συνιστοσών της Επιτροπής μας. Είστε υπέρ του αιτήματο αναβολής ε, το οποίο κατέθεσε η κυρία Ντάνοκα. Ο κύριος Τσίτσεστερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μίλησα προηγουμένως για το θέμα αυτό στην συνεδρία των συντονιστών, αλλά ευχαρίστω υποστηρίζω τις κυρίες Βέρτμαν και Σντάνοκα για την αναβολή του ε, θέματος. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής παρακαλώ ψηφίζουμε. Ποιοι είναι κατά. Εννέα ψήφοι κατά αποχές. Ευχαριστώ κύριε την πρόεδρος. Λοιπόν, δέκα κατά της αναβολής, 4 υπέρ της αναβολής, καμία αποχή, απορρίπτεται το αίτημα. Επιβεβαιούνται λοιπόν οι αποφάσεις ε, για την ημερήσια διάταξη ε, όπως ακριβώς έχουν προταθεί. Συνεχίζω με το τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έχει ο συνήθως διανεμηθεί το τμήμα Β με τις προτάσεις των αναφορών οι οποίες θα πρέπει να τερματιστούν. Έχει ήδη διανεμηθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση από πλευράς μου γύρω από αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Έχει κλείσει πλέον αυτό το τμήμα της ημερήσιας διάταξης και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο όπως ακριβώς ε, έχουμε ήδη ανακοινώσει και εγκρίνει είναι το σημείο 11 το σημείο 11 λοιπόν είναι η αναφορά 0338 του 12 του Γεωργίου Φλωρά, Έλλην πολίτης, για την εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του ανταγωνισμού από πλευράς της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχουμε εδώ ανάμεσά μας τον αναφερόμενο, έχει το λόγο για 5 λεπτά ο κύριος Φλόρας. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, το πρόβλημά μου με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κρατάει πολλά χρόνια. Άρχισε με την υποβολή ενός παραπώνου κατά του καρτέλ της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και των βιβλίων της. Αλλά υπήρξε η θελημένη καθυστέρηση για να ωφεληθεί το καρτέλ αυτό κατά των συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών που πληρώνουν υπερβολικές τιμές για τα διδακτικά βιβλία. Επίσης αναφέρθηκα στην Επιτροπή Αναφορών που πρώτη φορά έκρινε ότι είχα δίκιο το 2001. Τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2009 με τρομερή καθυστέρηση επέβαλε πρόστιμα 20 εκατομμυρίων ευρώ στα μέλη του καρτέλ και με δικαίωσε. Οχτώ χρόνια όμως κράτησε η διαδικασία. Είχα λοιπόν δίκιο που αναφέρθηκα, που παραπονέθηκα. Προσέφυγα στο δικαστήριο για την καθυστέρηση και η αναφορά δεν συμπεριλαμβάνει την τελική απόφαση. Τον Ιούνιο του 2013 ο Άριος Πάγος με απόφαση του με δικαίωσε με μια τελική απόφαση που προέβλεψε μεγάλη αποζημίωση για τις καθυστερήσεις. Γιατί εγώ επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ζημιωνόμουν. Δεν συζητάμε όμως αυτά σήμερα. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάει η Επιτροπή Αναφορών είναι ένα μικρό τμήμα της υπόθεσης αλλά πολύ σημαντικό. Σημαντικό διότι δίνει το δικαίωμα σε καρτέλ να προσφύγει χωρίς δικαίωμα στον ζημιονόμενο να κάνει το ίδιο. Τον Ιούλιο του 6 η Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι υπήρξε σύσταση καρτέλ για τα διδακτικά βιβλία ξένων γλωσσών. Αλλά η υπόθεση πάγωσε τελικά το 9 για λόγους που δεν εξηγήθηκαν. Δύο χρόνια μετά έγιναν νέες συστάσεις για την ίδια υπόθεση. Στη νέα σύσταση λοιπόν δεν υπάρχει πια η κατηγορία για σύσταση καρτέλ. Αυτό μας εξέπλησε. Μας εξέπληξε και μελετήσαμε την απόφαση και είδαμε ότι θεωρήθηκε <clears throat> ως ελαφρυντικό το ότι εστάλησαν επιστολές από την ε, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και αυτό θεωρήθηκε παρκές. Με βάση αυτές τις δηλώσεις οι επιστολές έδειχναν ότι υπήρχε επιθετική συμπεριφορά από δύο μέλη του καρτέλ. Αλλά αυτές οι επιστολές δεν μου εστάλησαν επισήμως και δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν αυθεντικές και δεν τις έγραψαν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, τα μέλη του καρτέλ δηλαδή. Κι όμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις δέχτηκε ως γνήσιες. Και έτσι αφαίρεσε τη σοβαρότερη κατηγορία της σύσταση καρτέλ. Το ξαναλέω για να είναι σαφές ότι τον Ιούλιο του 6 η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε καταδικάσει για σύσταση καρτέλ τους δύο πολιτές και επειδή βρήκαν στα συρτάρια τους μετά κάτι επιθετικές λέει επιστολές που τις υπέβαλαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αθωώθηκαν τελικά ενώ δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Τις δέχτηκαν ως γνήσιες τις επιστολές και γι' αυτό αφαίρεσαν την κατηγορία σύστασης καρτέλ. Και τώρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για κάτι τέτοιο. Αυτό έχει γίνει λοιπόν πια προηγούμενο και για άλλα καρτέλ οποιαδήποτε εταιρεία κατηγορείται για σύσταση καρτέλ μπορεί τώρα να δημιουργήσει πλαστά γράμματα, επιστολές χωρίς καμία απόδειξη γνησιότητας και αφαιρούνται οι κατηγορίες, αθωώνονται. Δεν ξέρω πώς μπόρεσαν να δεχτούν τέτοια στοιχεία. Και αφού τα δέχτηκαν θα τα δεχτούν και σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα σας διαβάσω 7 γραμμές για αυτά που είπε ο Υπουργός κ. Ξινίδης προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Βουλή. 4 Απριλίου 12 είναι στο φάκελο και ο κύριος Ξινίδης, ο Υφυπουργός, λέει στα ελληνικά. Κύριο Κυριτσάκη στην υπόθεση Φλωρά. Mr. Kiritsakis is the president of uh, the Greek Competition Committee. Πληθώρα ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουν φτάσει στα χέρια μου που αφορούν στο καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου. Κυρίω αφορούν την εκτίμηση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι δεν θεμελιωνόταν η ύπαρξη εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των εταιριών. Μπορείτε κύριε Σαλαβράκο να πείτε στον ομιλητή να μιλάει πιο αργά, δεν μπορούν να τον μεταφράσουν. και περιεχομένου. Δημιουργείται δηλαδή μια επικίνδυνη πρακτική. Ευχαριστούμε περίπτωση προσκόμιση επιστολών άνευ βεβαία ημερομηνία και περιεχομένου από επιχειρήσει που κατηγορούνται για καρτέλ, αυτέ θα απαλλάσσονται από τι κατηγορίε. Ουδέποτε υπήρξε επαρκή και αιτιολογημένη απάντηση του Προέδρου τη Επιτροπή στο θέμα αυτό. Mr. President, let's say that Floras is crazy. Is the... Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρελό ο Φλωρά, είναι και ο υφυπουργό ε, Τρελό. Φαίνεται ότι δεν ισχύουν στην Ελλάδα οι κανόνε του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ λοιπόν η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλούμαστε να εξετάσουμε ένα θέμα. Με ακούτε? Που θέτει ο αναφερόμενος και που έχει σχέση με την Εθνική Αρχή για τον Ανταγωνισμό, την Ελληνική Εθνική Αρχή αναφέρθηκε νομίζω ο αναφερόμενος και στον Γενικό Γραμματέα ή Υφυπουργό, τον Έλληνα, πάντως αυτό διευκρινίζω. Πρόκειται για υπόθεση εκπαιδευτικών βιβλίων σε ξένες γλώσσες που κρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2009. Ο αναφερόμενος ήταν ο προσφεύγων στην περίπτωση αυτή. Ο προσφεύγων λοιπόν υπήρξε επιτυχή στην περίπτωση αυτή. Η καταγγελία του οδήγησε σε έρευνα σε βάθος και κατέληξε σε δύο αποφάσεις επιβολής. Έκρινε η Εθνική Αρχή του Ανταγωνισμού ότι υπήρχε συλλογική δεσπόζουσα θέση των καθών, ότι κατεχράστηκαν την δεσπόζουσα θέση και σε ξεχωριστή απόφαση έκριναν ότι είχαν υπάρξει και κάθετοι περιορισμοί. Επομένω, πολύ σημαντικά πορίσματα και επιβλήθηκαν σημαντικά πρόστιμα στους καθών. Παρ' όλα αυτά, ο αναφερόμενος εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι δεν είναι ικανοποιημένο λόγω της εγκατάλειψης άλλου τμήματος της υποθέσεως, δηλαδή της concerted practice, που εγκαταλείφθηκε στην πορεία από τις αρχές και θεωρεί ότι η ελληνική εθνική αρχή δέχθηκε απαλλακτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι πολύ ελαφρά την καρδία και θεωρεί ότι ορισμένε από τι επιστολέ αυτέ ίσω να είναι και αναλυθεί. Απαντώντα, α υπογραμμίσω πρώτα, και το είπα και προηγουμένω, ότι η υπόθεση αυτή κρίθηκε από την Ελληνική Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού και επομένως και των ελληνικών εφετείων καθήκον ήταν να εξετάσουν την απόφαση και να δουν εάν συμμορφώνεται προς τον νόμο. Δεν είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε υπόθεση. Αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε προσφυγή και κατά των δύο αποφάσεων της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Τραγωνισμού και τα αρμόδια δικαστήρια τις επιβεβαίωσαν ωστόσο ο αναφερόμενος θα είχε την ευκαιρία ως προσφεύγων να συμμετάσχει στις δικαστικές διαδικασίες, αλλά από ό,τι, μαθαίνουμε επέλεξε να μην το πράξει. Ωστόσο, κατήγγειλε τις πρακτικές αυτές, έκανε και άλλες προσφυγές όπου είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του, ακολούθησε όλες τις δικαστικές οδούς και από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων στην Ελλάδα. Εμείς ως Κομισιόν οφείλουμε να το εξετάσουμε γενικότερα και να ρωτήσουμε είναι δυνατόν η συγκεκριμένη αυτή υπόθεση, η συγκεκριμένη αυτή πτυχή μιας υποθέσεως να αποτελέσει αιτία ανησυχίας για την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού και των δικαστηρίων. Εκεί πρέπει να βασίσουμε βέβαια την εξέτασή μας στα γεγονότα και βλέπουμε ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια λεπτομερής πτυχή μιας υποθέσεως, υποθέσεως η οποία πέρασε από τα δικαστήρια και επί της ουσίας της η απόφαση του πρώτου δικαστηρίου τηρήθηκε και από το ε, εφετείο. Ωστόσο, αυτά έχουμε επιτάπητος. Δεν έχουμε άλλες ενδείξεις και ούτε είναι προφανές ότι είναι γενικευμένο το θέμα. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι πάντοτε υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε υπόθεση ανταγωνισμού και οι καθόν επίσης βεβαίως έχουν το δικαίωμα να δικαστούν δίκαια και είναι γενικός κανόνας ότι καταρχήν η Εθνική Αρχή του Ανταγωνισμού φέρει το βάρος της αποδείξεως, να αποδείξει δηλαδή ότι υπήρξε παραβίαση. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τότε είναι σωστό να απαλλάξει από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Η νομολογία καθορίζει το επίπεδο των αποδείξεων και δεν ανησυχούμε εμεί ότι μπορεί να υπάρξει αρνητικό προηγούμενο γενικότερα δεν έχουμε και ενδείξει ότι η ελληνική αρχή ανταγωνισμού είναι, λαμβάνει πολύ ελαφρά υπόψη τα απαλλακτικά στοιχεία. Γνωρίζουμε, έχοντας έλθει σε επαφή, ότι η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού, η Ελληνική Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού, επιβάλλει τους κανόνες. Ήδη από το 2009, η Επίτροπος Κρούς, που ήταν τότε αρμοδία για τον ανταγωνισμό, έγραψε στην Επιτροπή σας ότι το ιστορικό επιβολής της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού είναι και παραπάνω από τον μέσον όρο κρατών μελών ε, παρόμοιου μεγέθους. Αυτό επιλέξει. Να μνημονεύσω ακόμη ότι τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας αναφέρονται σε υπόθεση του 2009. Εν τω μεταξύ έχει περάσει κάποιος χρόνος και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην ίδια την Ελλάδα για να ενισχυθεί το σύστημα επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού. Έχει γίνει λοιπόν αναθεώρηση και του σχετικού νόμου το 2011, καθώς επίσης έχει ενισχυθεί το προσωπικό της ε, αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού. Προσλήφθηκαν νέα πρόσωπα και η αρχή την οποία έχουμε μπροστά μας τώρα, στο ελληνικό πλαίσιο, είναι μια αρχή πολύ διαφορετική από αυτήν που ήταν το 2009. Εν ώψη του ιστορικού αυτού μας φαίνεται πολύ δύσκολο να αντλήσουμε ακόμη σήμερα συμπεράσματα από τα όσα συνέβησαν το 2009. Άλλωστε αυτά έχουν εξεταστεί ευρέως στα δικαστήρια. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι εμάς μας φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτή η υπόθεση. Ασφαλώς είναι ορθό να εξετάζει κανείς την, και στα προσεκτικά τις δραστηριότητες της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού. Αλλά από κάθε άποψη θεωρούμε ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει, να κλείσει την συγκεκριμένη υπόθεση και να αφιερώσει πλέον την προσοχή της στην διερεύνηση, εξέταση και αποκάλυψη άλλων υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ ευχαριστώ κύριο Σαλαβάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να πω και εγώ ότι πράγματι η αρχή ανταγωνισμού με τον νέο της Πρόεδρο τον κύριο Κυριτσάκη είναι πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν προηγούμενα. Ε, όμως εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη υπόθεση του 2009 κατά την οποία ο αναφέρον είχε προσφύγει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με δύο αιτήματα όπως προκύπτει από το φάκελο. Το ένα αίτημα αφορούσε την ε, ε, σύσταση κατά κάποιο τρόπο καρτέλ και το άλλο αίτημα είναι εκείνο για το οποίο δικαιώθηκε και επευλήθη στους ε, αντιπάλους του ένα σημαντικό πρόστιμο. Το θέμα για το οποίο παραπονείται από ό,τι μελέτησα είναι το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε καθοδόν ε, μια πράξη της Επιτροπής Συνταγωνισμού η οποία ήταν το κατηγορητήριο κατά των αντιπάλων εταιριών και έφυγε το στοιχείο της δημιουργίας καρτέλ. Εξηγήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι αυτό έγινε διότι υπήρξαν διάφορες επιστολές εκ των οποίων προέκυπτε ότι οι εταιρείε αυτές ή στο παρελθόν είχαν μεταξύ τους αντιπαλότητα και επομένω δεν είχαν συστήσει καρτέλ. Το πρόβλημα επομένω το οποίο γεννάται είναι εντελώς νομικό, θα κριθεί από τα δικαστήρια εάν και κατά πόσον οι λήψεις υπόψη ορισμένου εγγράφου πρέπει να γίνεται μια ορισμένη διαδικασία διότι ο νόμος στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη προβλέπει με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται από τα δικαστήρια ή από τις αρχές οι οποίες ε, απονέμουν ε, στις οποίες έχει απονεμηθεί η ιονή δικαστική διαδικασία ε, οι λήψεις αποδεικτικών στοιχείων. Φαίνεται ότι εδώ παρεδιάστη ο τρόπος εξ όσων γνωρίζω και σαν νομικός ε, ε, έχω αντίληψη των ελληνικών πραγμάτων φαίνεται παρεβιάστη ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη έγγραφα και αυτό προφανώς οφείλεται σε συγκεκριμένους υπαλλήλου της γραμματείας ε, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν προκύπτει εάν είναι γενικευμένη αυτή η πρακτική. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια εκκρεμής δικαστική διένεξη από ό,τι είδα στο φάκελο και υπάρχει μια δικαίωση του προσφεύγοντος από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο τον δικαιώνει ως προς το θέμα της καθυστέρησης λήψεως αποφάσεων και του επιβάλλει για ηθική βλάβη στο ελληνικό δημόσιο υπέρ του προσφεύγοντος το ποσό των 350.000 ευρώ το οποίο είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό ποσό βεβαίως ποσών αποζημιώσεως διαθηκιούδανα. Κατά τις αποφάσεις αυτής όμως του διοικητικού εφετείου, η οποία είναι πρόσφατα, του 2013, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο High Court δηλαδή. Επομένως, αναμένεται οριστική απόφαση, τελε, αμετάκλητη απόφαση, διότι αυτή είναι τελεσίδικη μόνο, από το High Court εντός των προσεχών ημερών, ε, μηνών. Ε, γι' αυτό θα έλεγα ότι θα μπορούσε να μείνει ανοιχτή η ε, αναφορά, να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου και να δούμε εάν πέραν της αποφάσεως αυτού του ελληνικού δικαστηρίου γίνονται σκέψεις για παραβίαση των αρχών για τις οποίες ενάγει την Επιτροπή Ανταγωνισμού ο ε, παριστάμενος εδώ αναφέρον. Συνιστώ λοιπόν να κρατηθεί ανοιχτή. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαβράκο. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφού άκουσα τον αναφέροντα ή αναφερόμενο και την Κομισιόν, βλέπω ότι είναι μια περίπτωση υπερβολικής καθυστέρησης. Δεύτερον, αν ένα ελληνικό δικαστήριο με τα στοιχεία που διαθέτει αποφασίσει ότι υπήρξε παραβίαση και επιβεβαιώσει ότι υπήρχε ένα είδος καρτέλ όχι των μεγάλων βιομηχανιών για υποβρύχια και αεροπλάνα αλλά για βιβλία ξένων γλωσσών τι άλλο χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε ότι η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τον ανταγωνισμό δεν έγινε σωστά, για να μην πω. Για να μην λάβω υπόψη με αυτά που μας είπε ο κύριος Σαλαβράκος, δηλαδή ότι μπορεί οι υπάλληλοι της αρχής ανταγωνισμού στην Ελλάδα μπορεί να είχαν διαρρεύσει στοιχεία της υπόθεσης και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι η σωστή εφαρμογή του νόμου και σωστή συμπεριφορά μιας αρχής που στοχεύει στην ε, σωστή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Εγώ νομίζω ότι όχι. Και αυτό δεν είμαι ικανοποιημένο από την απάντηση της Κομισιόν που μας λέει ότι η Ελλάδα έχει υψηλότερα πρότυπα και από άλλες χώρες μέλη. Όχι, αν, αν έχει υπάρξει παραβίαση που την έχει επιβεβαιώσει και δικαστήριο, τότε είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μάλιστα όχι στο βασίλειο της Δανημαρκίας, αλλά στην Ελλάδα. Άρα καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι. Τέλος. Μετά από τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια λέγω, θα κλείσει μάλλον τελικά η υπόθεση, αλλά γιατί η Κομισιόν δεν επιτηρεί σωστά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη την ενωσιακή νομοθεσία και όχι μόνο για τον ανταγωνισμό συνήθως μας λένε το ίδιο συμβαίνει και για το περιβάλλον και για άλλα θέματα, αλλά δεν έχουμε προσωπικό για να επιτύχει. Θυμάμαι ότι όταν πρόκειται για θέματα μεγάλων επιχειρήσεων ή πολυεθνικών, συνήθως η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προσέχει περισσότερο τα πράγματα, αντιδράει πολύ γρηγορότερα και η εταιρεία που έχει ζημιωθεί από την απόφαση της αρχής ανταγωνισμού συνήθως δικαιώνεται από την Κομισιόν. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί εδώ πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις. Τα βιβλία δεν είναι κανένα θέμα τεραστίων συμφερόντων, είναι μικρές επιχειρήσεις. Άρα μια παραβίαση που συμβαίνει εδώ θα επαναληφθεί και για σπουδαιότερα θέματα. Τώρα μας λένε δεν υπήρξε καρτέλ. Αν όμως δεν υπήρξε καρτέλ, στην περίπτωση αυτή, τότε οι δύο εταιρείες που συμπεριφέρθηκαν έτσι μονοπωλιακά το έκαναν αυθορμήτως με ποια βάση σε ποια βάση Βεβαίω και ήταν σύσταση καρτέλ. Έτσι έδρασαν ως καρτέλ. Πρέπει λοιπόν η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και ελπίζω την επόμενη φορά η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να μας δώσει πολύ πιο σοβαρά συμπεράσματα. Αφού έχουμε δικαστική απόφαση που λέει ότι υπήρξε παραβίαση, ήταν λάθος, και επιβλήθηκε κύρο, κύρωση. Αν δεν αρκούν οι κυρώσεις και τα πρόστιμα, τι αρκεί. Κύριε Γιάρη, θα συμπληρώσω αυτά που είπαν οι δύο συνάδελφοί μου και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά και άλλωστε να πρόκειται σε εμά την Επιτροπή Αναφορών να επανεξετάσουμε την αναφορά αυτή πριν από το πέρας τη κοινοβουλευτική περίοδου. Συμφωνώ δε στα υπόλοιπα με τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι συναδελφοί μου. Εκ νέου ο λόγος στον αναφέροντα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευγενική για τα χρόνια πριν το 2009. Οι λέξεις ήταν πολύ προσεκτικά βαλμένες. Σήμερα λέει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Προφανώ όμω η Επιτροπή δεν αγοράζει προϊόντα από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ του Βελγίου. Γιατί θα ήξερε ότι είναι, έχουμε τα πιο ακριβά προϊόντα σε σχέση με τα εισοδήματά μα στην Ελλάδα. Μίλησε για διαφορετικά πρόσωπα. Το φάουλ αυτό, κυρία Πρόεδρε, που έγινε το 2006 και το 2008, το έκανε το ίδιο πρόσωπο σαν Διευθύντρια Νομική Υπηρεσία, που είναι σήμερα η Γενική Διευθύντρια τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα τα πρόσωπα δεν αλλάξανε, παραμένουν τα ίδια. Αν μια πρακτική που έγινε τότε είναι φάουλ, θα είναι φάουλ και στο μέλλον. Ε, είπε η Κομισιόν ότι εξετάστηκε στα δικαστήρια τα οποία συμφωνήσανε με την απόφαση. Θα ήθελα να πληροφορήσω την Κομισιόν ότι η εναρμονισμένη πρακτική που αφαιρέθηκε δεν εξετάστηκε στα δικαστήρια γιατί δεν υπήρξε εισήγηση για να την εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό ήταν το δώρο που κάνανε σε αυτές τις εταιρείε. Ε, η Κομισιόν τελικά όμως δεν απαντάει. Αυτή η συγκεκριμένη πρακτική, εγώ δεν ήρθα σήμερα εδώ να μιλήσω για 10 χρόνια που μαλώνω με τα καρτέλ και την Επιτροπή. Αυτή η συγκεκριμένη πρακτική την αποδέχεται να μπορεί να φέρει ένα καρτέλ, αν τη φέρει αύριο μια κατηγορούμενη εταιρεία εδώ, αφού έχει βγάλει εισήγηση, λευκές επιστολές, θα τις δεχτεί η Κομισιόν σαν αποδεικτικό στοιχείο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ είμαι πρόεδρο στην Επιτροπή για θέματα ανταγωνισμού στο μεγαλύτερο επιμελητήριο τη Ελλάδο. Έχουμε 160.000 μέλη. Γνωρίζω πολύ καλά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ποτέ η Κομισιόν δεν κάλεσε κάποιον από εμά να του πούμε τι γίνεται. Τα καρτέλ είναι πανίσχυρε εταιρείε που αδιαφορούν για το διασυρμό. Του απασχολεί μόνο οι αστικέ και ποινικέ ευθύνε και τα πρόστιμα. Και γνωρίζουμε όλοι, κυρία Πρόεδρε, ότι από μία λεπτομέρεια αλλάζουν όλα. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι το βασίλειο των καρτέλ. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ λοιπόν επί τη βάση αυτών που ακούσαμε από τον αναφέροντα και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα αιτήματα των μελών που πήραν το λόγο θεωρώ ότι θα ήταν πιο εύθετο να μείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά και να ζητήσουμε κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις, πιθανώς γραπτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προσποθήσουμε να βγάλουμε την υπόθεση από αυτό το πεδίο αβεβαιότητας το οποίο είναι βυθισμένη και να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των ερευνών ε, τις οποίες έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικά επίσης με την επιλογή ε, των συνομιλητών που θα μας ενημερώσουν για το εάν ε, τα επιχειρήματα που ακούστηκαν είναι τεκμηριωμένα ή όχι. Καλό λοιπόν να διευκρινίσουμε τα πράγματα καλύτερα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει μια λεπτομερέστερη γραπτή απάντηση και θα αποφασίσουμε από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε ανάλογα με το περιεχόμενο της απάντησης αυτής. Ευχαριστώ τον αναφέροντα που ήταν ανάμεσά μας και παρουσίασε την αναφορά του. Και περνώ τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ε, ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε. Είναι το σημείο 6, η συζήτηση δηλαδή για την έκθεση για την αποστολή στην Γαλλικία της Ισπανίας. Ο κύριος Μπουλάν έχει ζητήσει το λόγο. Okay, one minute to Α, ωραία, κυρία Στανόκα, διαδικαστικό. Θέλω να κάνω μία δήλωση. Δεν είμαι σε θέση να συμμετάσχω στη συζήτηση των τροπολογιών διότι δεν μεταφράστηκαν σε γλώσσες που καταλαβαίνω. discuss the amendment. Και δεν είναι δυνατόν να τη συζητάμε όταν εμείς τα δύο μέλη της τριμελούς αποστολής των, των τριών υπευθύνων για το περιγραφικό μέρος δηλαδή διαφωνούν με το περιγραφικό αυτό μέρος που έχει υποβληθεί. Υπάρχει εδώ μια συνωμοσία των μεγάλων πολιτικών ομάδων για να εγκριθεί η έκθεση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την θέση των δύο από τα τρία μέλη της αποστολής. Φυσικά μπορούμε να ψηφίσουμε και με τη μηχανή ακόμα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω σε τέτοια παιχνίδια και θα γράψω σήμερα επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να εξηγήσω πώς διεκπεραιώνεται η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ κυρία Σντάνοκα. Λυπάμαι που εγκαταλείπετε. Λυπάμαι που δεν συμμερίζεστε την λογική που λέει ότι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απόφασης προς όφελος των πολιτών θα πρέπει να αντικαταστήσουμε ε, την έλλειψη απόφασης με την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής της ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπουλάν. Μη μακρηγορήσετε παρακαλώ. Ε, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν χαίρομαι για την σοφή απόφαση της Επιτροπής μας που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε για να καταπολεμήσουμε τις δημόσιες ή όχι και τόσο δημόσιες προσπάθειες παρεμπόδισης του έργου μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ενώπιον των πολιτών της Ισπανίας και της Γαλλικίας ιδιαίτερα αλλά και γενικότερα των Ευρωπαίων. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, ευχαριστώ τους συναδέλφους που τις κατέθεσαν, υπάρχουν 84. Οι περισσότερες στα ισπανικά. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι χάρη στο νέο εργαλείο μετάφρασης που έχουμε τώρα στο Κοινοβούλιο Πάρα πολύ γρήγορα έχουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες όλων των κειμένων ακόμη και στα ισπανικά. Και χάρη σε αυτό μπόρεσα να εξετάσω τις τροπολογίες και να μιλήσουμε σήμερα για αυτές. Θέλω να τονίσω μερικά στοιχεία. Η τροπολογία 1 μου φαίνεται απαράδεκτη λόγω του άρθρου 167β που ζητάει αντικατάσταση ενός κειμένου από άλλο. Εσείς κυρία Πρόεδρε θα δείτε αν είναι αποδεκτή ή όχι. Εγώ όμως θέλω να ήθελα να δηλώσω ότι πρόκειται για νέα προσπάθεια καθυστέρησης. Δεύτερον, έχουν κατατεθεί τροπολογίες εξ ονόματος κάποιου που δεν είναι πια ευρωβουλευτής. Αν κάποιος θέλει να τις αναλάβει μπορεί να το πράξει αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να αναφέρουμε το όνομα ενός τρίτου που δεν είναι πια ευρωβουλευτής. Δεν ζητώ να θεωρηθούν απαράδεκτες, είναι σωστές και αποδεκτές και πρέπει να τις ψηφίσουμε, αλλά να φύγει από αυτές το όνομα του πρώην Ευρωβουλευτού. Έπειτα, θέλω να προσέξετε ότι απαράδεκτες είναι και άλλες τροπολογίες που αναφέρονται σε μη αποδεκτές αναφορές ή σε αναφορές που μιλούν για τη Ρία Ντεφερόλ και που πρέπει να θεωρηθούν μία αποδεκτές. Είναι η τροπολογία 4, 5, 10 και 59. Ας μην επισέλθω στις λεπτομέρειες του θέματος γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά. και θα χρειαζόταν πολλής χρόνος, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τις τροπολογίες. Οι περισσότερες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και αποδεκτές του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών, της ΓΚΟΕ και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ε, Mrs κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για το παραδεκτό ή μη παραδεκτό αιτήματο να καθόμαστε να συζητούμε αιτήματο το οποίο είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι είναι περιττό. Άλλωστε ούτε θέλω να μπω στην ουσία του θέματος. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου μονάχα για μια προσπάθεια του συναδέλφου να περάσει άλλη μια φορά με το ζόρι την θέση του. Μα είχε πει και τότε, είμαι επικεφαλή αντιπροσωπεία και πρέπει να κάνετε ό,τι λέω. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Για τι άλλε τροπολογίε έχω να πω μόνο ότι κατανοώ βέβαια την ισπανική γλώσσα, αλλά όχι τόσο καλά. Δεν τι καταλαβαίνω όλε τι λεπτομέρειε. Γι' αυτό θα ήθελα τουλάχιστον να έχουμε την αγγλική μετάφραση των ισπανικών κειμένων. Και γι' αυτό ε, παρακαλώ αυτό να ληφθεί υπόψη. Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορώ ωστόσο να τα κατανοήσω όλα. Τις υπόλοιπες συζητήσεις μπορούμε και να τις αφήσουμε, δεν χρειάζεται να τις κάνουμε, τις κάναμε χθε. Νομίζω ότι οι τροπολογίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και καλές και ασφαλώς θα υποστηρίξω ορισμένες τροπολογίες συναδέλφων μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. Επανήλθαμε στο θέμα των τροπολογιών. Εδώ είχαμε συμφωνήσει για το χρονοδιάγραμμα. Οι τροπολογίες ε, είναι στο στάδιο της μετάφρασης. Δεν θα ψηφιστούν σήμερα, γιατί οι συνάδελφοι δεν είχαν την δυνατότητα τουλάχιστον στα αγγλικά να τις έχουν στη διάθεσή τους. Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, δεν πρέπει να ανησυχείτε ως προς το θέμα της μετάφρασης. Στην παρούσα φάση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε της γνώσης αυτών που δεν πήραν μέρος επί τη βάση της εκθέσεως και επί τη βάση των τροπολογιών οι οποίες έχουν κατατεθεί και τις οποίες κάποιοι ή τις περισσότερες γνωρίζουμε. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία θα είναι όλοι ενήμεροι σε βάθος για το περιεχόμενο των τροπολογιών. Μιλαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής δεν θα πρέπει να επιτρέψει να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες να δεσμεύουν την λήψη αποφάσεων. Έχουν υπάρξει προσπάθειες παρεμπόδισης της διαδικασίας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι με τις ε, συγκεκριμένες αποφάσεις θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα για τη βελτίωση ε, της κατάστασης ε, στην συγκεκριμένη περιοχή και θα ζητήσουμε από τις τοπικές αρχές και στον τομέα των καθορισμών των υδάτων να φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τους τις ανηλυμένες σχετικά με τον κοινοτικό νόμο. Κάποιες από τις τροπολογίες που καταθέσαμε μαζί με τον Ιτουργκάιθ είναι γλωσσικές. Ε, ε, θα πρέπει να ονομάζεται σωστά το συγκεκριμένο μικρό ποτάμι, ε, γιατί δεν διευκρινίζεται στην έκθεση. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, τροπολογίες που διευκρινίζουν λίγο καλύτερα το κείμενο. Κάποιες άλλες έχουν μεγαλύτερο βάρος και προσπαθούν να αλλάξουν κάποιες συγκεκριμένες φράσεις. Πάντως, είναι θετικό το ότι καταλήγουμε πλέον. Ε, νομίζω ότι οι τροπολογίες μας και του κυρίου Ιτουργκάιθ είναι τροπολογίες επικοδομητικές. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα προτινόμενα και να διευκολύνουμε επιτέλους η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάει στις περιφερειακές αρχές και να κρατήσουμε τα μικρά αυτά ποτάμια καθαρά. Thank you. Ευχαριστούμε. Α, καλά, εσείς με το δύσκολο όνομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρόκειται για μια έκθεση, έχει περάσει από πάρα πολλά και πράγματι ο δρόμος που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα ήταν στρεβλός. Άκουσα τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Στάνοκα και ε, Βέρκμαν και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε πολλά μαζί τους. Όταν έχεις να εξετάσεις τροπολογίες και δεν γνωρίζεις τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες, αυτό δεν είναι δημοκρατικό και διαφανές και δικαιολογείται η αντίδρασή τους. Για τον κύριο Μπουλάν, πριν έρθω σε αυτό το κοινοβούλιο εγώ είχα ασχοληθεί με θέματα που άπτονται της αυτόματης μετάφρασης και τα λοιπά, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τι ε, προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η αυτόματη μηχανική μετάφραση σε τέτοιου είδους κείμενα. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, το κόμμα, η τελεία, ο τόνος και σε αυτή την περίπτωση η αυτόματη μηχανική μετάφραση δεν είναι ε, καθόλου ικανοποιητική. Τώρα, για την ουσία της υπόθεσης. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή ε, ε, σημειώνει την διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας και τα δύο μέλη της αποστολής του. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή δεν αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία οι αναφέροντες ε, ε, μας έχουν ε, δηλώσει και σε μας και στην Επιτροπή. Το θέμα της κατάστασης των ποταμών της Γαλλικίας είναι ένα σημαντικό θέμα και μέσω των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και από ε, τις άλλες τροπολογίες φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται με πάρα πολύ μικρή ταχύτητα και δεν εφαρμόζεται σωστά μέχρι τώρα η κοινοτική νομοθεσία. Ε, θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ε, τα κείμενά μας την πραγματικότητα της κατάστασης στο σύστημα αυτό των ποταμών της Γαλλικίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε σαν Επιτροπή και υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες ε, τις οποίες έχει καταθέσει ο κύριος Μέγερ ε, που δίνουν πραγματικά ε, την κατάσταση ως έχει γιατί αλλιώς η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση light με γλυκαντικές ουσίες που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ευχαριστώ εγώ την Προεδρία για την προσπάθεια την οποία έκανε για να ολοκληρωθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ συμφωνώ και με το περιεχόμενο της παρουσίασης του κυρίου Μπουλάν και με το περιγραφικό τμήμα με το οποίο διαφωνούν οι δύο συμμετέχουσες βέβαια στην αποστολή και που δεν μας έδωσαν μια πραγματικά εναλλακτική ε, περιγραφή, απλά ε, το θέμα δεν είναι οι απόψεις προσωπικά όλου των ενδιαφερομένων, αλλά οι απόψεις αυτών που πραγματικά ήταν επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας θα πρέπει λοιπόν το κείμενο αυτό να περιελάμβανε τις απόψεις όλων όσων πήραν μέρος, ιδιαίτερα σε σχέση με τα τμήματα τα οποία δείχνουν τα, ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να αποκτήσουν κίνητρα και οι ισπανικές αρχές σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν. Δημιουργείται μια καθυστέρηση με αυτό το οποίο συνέβη μέχρι τώρα και αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουν κάνει οι αναφέροντες ασκούν τα δικαιώματά τους και ε, προσφεύγοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητούν μια απάντηση στα προβλήματα τα οποία θέτουν. Δεύτερον, και αυτό κάνουν οι τροπολογίες μου, ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν τον κοινοτικό κανόνα. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Θα πρέπει, σημειώνοντας την καθυστέρηση η οποία έχει υπάρξει, να προσπαθήσουμε να την καλύψουμε, αλλά να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι ε, πρέπει να υπάρξει πρόοδος, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αναφερόντων Θα πρέπει να αναδοθεί λοιπόν προτεραιότητα στις τοπολογίες οι οποίες βοηθούν στο να καλυφθεί η καθυστέρηση. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές της Ισπανίας από άλλες άλλων κρατών μελών. Ε, δεν πρέπει, ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σεβόμαστε γενικότερα τις δημοκρατικές αρχές. Είμαι υπέρ λοιπόν της διαφάνειας χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνολογούμε. Η Ισπανία είναι μια χώρα όπου υπάρχουν εγγυήσεις στον τομέα της παραγωγής των τροφίμων, στον τομέα των κτηνιατρικών ελέγχων. Υπάρχουν πάντα κάποια προβλήματα και μπορεί να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια και αναγνώριση όμως ταυτόχρονα ότι η Ισπανία είναι μια χώρα με επαρκείς ελέγχους και συνεπώς όλες οι ε, τροπολογίες οι οποίες τίνουν στην βελτίωση ε, της διαφάνειας πρέπει να γίνουν δεκτές. Σχετικά με την εταιρεία Ρεγκανόζα εμείς ε, νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και να δεχθούμε τις απαντήσεις τις οποίες μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει διάλογος ανάμεσα στην ε, επιχείρηση τη συγκεκριμένη και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Ε, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι στη διάθεση του συνόλου της κοινωνίας. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών να είναι προσβάσιμα σε όλους. Ε, μιλάμε για μία περίοδο κρίσης στην παρούσα φάση, υπάρχουν ε, περικοπές στον τομέα και της εκπαίδευσης και της υγείας, θα πρέπει τα μέτρα αυτά όμως για την ασφάλεια των καταναλωτών να συνεχίσουν να λαμβάνονται ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πω ότι για τις εγκαταστάσεις αυτές ε, μετά από τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε και με τους αναφέροντες και με τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης περιοχής και των εγκαταστάσεων θα πρέπει να δώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να κατανοήσουμε την κατάσταση του συγκεκριμένου αυτού πόταμου Εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κάναμε αυτό που έπρεπε απέναντι στους αναφέροντες. Μήνες μετά από τη συζήτηση της αναφοράς συνεχίζουμε να συζητάμε και είναι απαράδεκτο μια αποστολή ε, η οποία περιλαμβάνει τρία μέλη να μην είναι σε θέση να διατυπώσει μια συγκεκριμένη έκθεση με σωστό τρόπο. Η έκθεση την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος της αποστολής τη συγκεκριμένη της Επιτροπής μας δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των απόψεων των υπολείπων μελών, δηλαδή της πλειοψηφίας της αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τους ε, αναφέροντες. Εδώ θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Νομίζω ότι δεν θα ε, να αγνοήσουμε πλήρως και να περιφρονήσουμε τις συγκεκριμένες αναφορές. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία αποστολή η οποία δίνει ε, την εικόνα ότι δύο μέλη έχουν μία άποψη, ένα μέλος έχει μία άλλη άποψη και η άποψη του ενός μέλους είναι αυτή η οποία κυριαρχεί και τι λέει η άποψη του ε, προεδρεύοντος της Επιτροπής, του υπευθύνου αν θέλετε, ότι αυτά τα οποία γίνονται εκεί είναι όλα σωστά, ότι η κυβέρνηση η τοπική κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει και δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ε, λάθος, είναι κακό, δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, θα έπρεπε η αποστολή ή η εκθεση για την αποστολή να αντικατοπτρίζει το τι πραγματικά ε, ε, συμβαίνει και ποια είναι εν πάση περιπτώσει η άποψη της πλειοψηφίας. Και αυτό θα έπρεπε να γίνεται και να ολοκληρώνεται η διαδικασία ένα μήνα μετά και όχι δέκα μήνες αργότερα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη το να εξακολουθούμε τώρα να συζητάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά την συμβατότητα των μέτρων ε, της ε, βιομηχανικής εγκατάστασης με τα μέτρα και τους κανόνες για την προστασία της φύσης κτλ. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Εγώ είμαι αλληλέγγυος ε, με τις συναδέλφους Βέρτμαν και Σντάνοκα γιατί πράγματι ε, δεν έχει νόημα το συγκεκριμένο αυτό κείμενο το οποίο συζητάμε. θα έπρεπε να, πάμε, να στείλουμε μόνο του τότε τον κύριο Μπουλάν. Δεν είχε νόημα αυτό το οποίο έγινε, να πάει μόνος του να γυρίσει να μας κάνει την έκθεσή του και να μην χάσουμε την ουσία αλλά και τον χρόνο τον οποίο χάσαμε. Δεν θα πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο λοιπόν. Λέτε ότι η επιχείρηση αυτή έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγγυήσει για να λειτουργεί κτλ. Αν και είναι σχετικά κοντά λέει σε κάποιες κατοικίες, ε, σχετικά κοντά. Τι θα πει αυτό τώρα να μην κοροϊδεύουμε παρακαλώ. Είναι κολλητά πάνω, εν πάση περιπτώσει, στην βιομηχανική εγκατάσταση. Και η διατύπωση την οποία έχετε στην παρουσίασή σας, στην έκθεσή σας με εκπλήσει. Και μιλάτε για κάποια μέλη της Επιτροπής, όταν η κατά πλειοψηφία η αποστολή που ε, στείλαμε εκεί λέει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και όχι κάποια μέλη. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση λοιπόν, λυπάμαι γι' αυτό εγώ ζητώ συγνώμη από τους αναφέροντες. Εμείς δεν εγκρίνουμε τις μεθόδους που οι οποίες χρησιμοποιήσαμε, δεν μας αφορά η μέθοδος που ακολουθήθηκε, είναι αντιδημοκρατική η μέθοδος και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα στανούμε ε, ικανοί να παίρνουμε αποφάσεις με δημοκρατικό τρόπο. Η αλήθεια θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ε, ε, έκθεση και οι συστάσεις που γίνονται θα πρέπει να είναι ικανές να βοηθήσουν να λυθούν τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν αυτό το στόχο. Εγώ αμφιβάλλω βέβαια αν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Σίτουργκάης. Ευχαριστώ μετά την παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος Μέγερ θα μου επιτρέψει να του θυμίσω όπως και στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας ότι οι ισχυρισμοί των κυρίων, κυριών μάλλον Βέρτμαν και Σδάνοκα και τα σχόλιά τους ε, ελήφθησαν υπόψη από την πρόεδρό μας την κυρία Ματσόνη όταν ε, μας έστειλε το πρώτο κείμενο στην Επιτροπή. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι η κυριαρχία της δημοκρατίας και ο σεβασμός της δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο προβλέπει ο κανονισμός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και η κυρίαρχη στην Επιτροπή μας είναι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας τα τρία τέταρτα και πάνω από τα τρία τέταρτα αυτού του κοινοβουλίου. Ναι κυρία Βέρμαν έτσι είναι τα πράγματα, τα τρία τέταρτα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν οι φιλελεύθεροι ακριβώς τι απόψεις έχουν, δεν ξέρω ποια ήταν η στάση τους και σας άφησαν στην πολιτική σας ομάδα μόνοι, αλλά η πλειοψηφία μίλησε και να πω και στους άλλους συναδέλφους, ιδιαίτερα στον συνάδελφο που δεν γνωρίζω και είναι νέος στην συγκεκριμένη επιτροπή. Ε, να πω ότι δεν είναι υπεύθυνο ο κύριος Μπουλάν για το ότι δεν υπάρχουν α, μεταφράσεις, προσπάθησε να βρει μια άλλη λύση. Ε, έκανε ο κύριος Μπουλάν για να προσπαθήσει να καταλάβει. Είναι σαφές ότι οι μεταφράσεις οι οποίες γίνονται με μηχανικό, με αυτόματο τρόπο μέσω του διαδικτύου κτλ δεν είναι ε, απόλυτα έγκυρες. Αλλά να του αναγνωρίσουμε παρακαλώ την προσπάθεια την οποία έκανε και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα η γραμματεία μπορεί να εξηγήσει ή να εξηγήσει έστω και για το ότι δεν είναι ακόμα έτοιμες οι μεταφράσεις. Τελειώνοντας λοιπόν να κάνω ένα επιπλέον σχόλιο για το θέμα των τροπολογιών που ε, παρουσίασε η κυρία, που κατέθεσε η κυρία Μιράντα. που δεν είναι πλέον ε, ε, βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι κύριοι Μιλαν Μόντο και οι Τουργάιζ έχουν επίσης καταθέσει μια τροπολογία την 24 η οποία λέει εδώ έχει τα ονόματά τους ε, και του Φερνάντες Αλμπόρ που ήταν εδώ ε, είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο αλλά έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που έχει φύγει λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό και θα πρέπει να ε, τεθεί το θέμα και προς την γραμματεία να μας επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέγω εγώ τώρα σε σχέση με το αποδεκτό αυτής της τροπολογίας. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένες οι πλειοψηφίες που διαμορφώνονται κύριε Μέγερ και οι πλειοψηφίες αυτές καθιστούν κυρίαρχη την Επιτροπή μας και δείχνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οι οποίες έγιναν μέσω της Προεδρίας μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ιτουργκάης. Πριν περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο, γιατί ήδη έχουν οι συνάδελφοι αρχίσει το λόγο, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο και μετά θα συνεχίσουμε. What Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα έχουμε, θα έχουμε καταλήξει σε κάποια, σε συμπεράσματα και σε κάποιες συστάσεις. Στην παρούσα φάση θα ήταν πρόωρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τις θέσεις της Σημειώνουμε με ικανοποίηση τη διαδικασία στην οποία βρίσκεται η έκθεση γιατί υπογραμμίζει τα προβλήματα συγκεκριμένα μόλυνσης στα ποτάμια της περιοχής της Γαλλικίας ε, και που υπογραμμίζουν τα μέτρα αυτά τα οποία καλούμεθα να πάρουμε την μεγάλη σημασία που έχουν οι δυνατότητες νομικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν μπορούμε να επιφυλασσόμεθα κατά τα άλλα περιμένοντας το τελικό κείμενο από πλευρά σας. Thank you. Mrs. κυρία Βέρτμαν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επανέρχομαι σε αυτό το επιχείρημα περί δημοκρατίας. Έχει δίκιο ο Βίλι Μέγερ όσο και μεγάλη απόσταση να έχουμε πολιτικά, αλλά σε αυτό που είπε έχει δίκιο. Είναι αντιδημοκρατικό όταν έχω μια αντιπροσωπεία τριμελή, δύο από τα μέλη αυτά καταλήγουν σε μια απόφαση και ένα, το ένα μέλος που μένει δεν συμφωνεί. Αυτό λοιπόν λέω τότε, αυτή η μεμονωμένη άποψη έρχεται και μας λέει ότι αυτή θα ισχύσει. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Ο ρόλος της αντιπροσωπείας αμφισβητείται. Ήμασταν τρία μέλη. Εάν η άποψη, οι εντυπώσεις, οι εμπειρίες των δύο από τα τρία μέλη δεν μετρούν, τότε εγώ ισχυρίζομαι και θα το θέσω υπόψη και των συντονιστών, ότι πρέπει να καθίσουμε να ξανασκεφτούμε τον ρόλο αντιπροσωπιών που αποτελούνται παραπάνω από ένα μέλη. Όταν μονάχα μια άποψη, ένα έγγραφο και μόνο οι απόψεις του επικεφαλής της αντιπροσωπείας ισχύουν. Πολλοί με γνωρίζετε και από άλλες αντιπροσωπείες. Μπορούν τα πράγματα να γίνουν και διαφορετικά. Και βέβαια ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας λαμβάνει ορισμένες... Βίκτορ, σε παρακαλώ, μπορείς να τηλεφωνήσεις έξω από την αίθουσα. Ωστόσο, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε από κοινού του επικεφαλής και των μελών. Αυτή είναι η δική μου άποψη περί δημοκρατίας. Τι θέλουμε τη δημοκρατία με τις αποφάσεις της πλειοψηφία, εάν οι απόψεις πλειοψηφία δεν λαμβάνονται υπόψη. Θέλω και αυτό να συζητηθεί, ίσως όχι εδώ και τώρα διότι δεν έχουμε χρόνο, όλα αυτά θέλω να το θέσω επιτάπητος και να συζητηθεί. Κάρλος, μίλησες για την ψηφοφορία. Ψήφι 10 υπέρ, 4 κατά. Η ανάποδα. Πάντως, αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι τουλάχιστον τέσσερις έφυγαν. Ήταν λίγα λεπτά εδώ για να ψηφίσουν. Ναι εντάξει σύμφωνοι, προσήλθαν κάποιοι εδώ, ψήφισαν και απεχώρησαν. Είναι σωστό όμως να μην μπορούμε να πείσουμε τα πλήρη μέλη μας, τα τακτικά μέλη μας να ε, καθίσουν να ψηφίσουν και έρχονται οι αναπληρωτές και μετά φεύγουν ίσως πρέπει να την κλείσουμε κάποια στιγμή την Επιτροπή Αναφορών, διότι και εγώ θα μπορούσα να είχα φέρει στο κάτω της γραφής οποιουσδήποτε εδώ για να πω τώρα σηκώστε το χέρι σας για να ψηφίσουμε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να φέρνω κάποιον να ψηφίζει εδώ που δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται. Και αυτό θέλω να σας το θέσω υπόψη λοιπόν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να μας προβληματίσουν εδώ. Και last but not least που δεν το έχω συζητήσει ακόμη με την κυρία Σντάνοκα αλλά το θέτω και αυτό επιτάπητο το ερώτημα δηλαδή η πρόεδρος μας, άλλωστε το έτσι αποφάσισε, είμαστε υποχρεωμένες να το δεχτούμε, ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας επιβάλλεται, αλλά θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Εάν το έγγραφο, η γνωμοδότηση δηλαδή της Ντάνοκα και η δικιά μου, αν δεν μπορούν να μπουν ως δίθεν minority report και να προσαρτηθούν στην έκθεση ως έκθεση της μειοψηφίας, διότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο όταν ε, υποβάλλουν έγγραφο δύο μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας, το έγγραφό τους να γνωρείται. Ο Πρόεδρεύων. να πάτε στους, ε, και να πείτε στους ε, συναδέλφους σας και να τους πείτε όχι να έρθουν να ψηφίσουν αλλά και να εργάζονται κιόλας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ εσύ είσαι πάρα πολύ επιμελής, άλλους δεν τους βλέπω. Από τη δική μου ομάδα βλέπω, από άλλες ομάδες ναι. Από την ομάδα των φιλελευθέρων όχι. Πέστε τους λοιπόν, εμψυχώστε τους να έρχονται να ψηφίζουν. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, μου λέει ο γραμματέας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ποστινάρου, μετά Μέγερ και μετά Μπουλάν. Και παρακαλώ όλες και όλους, α και εσείς ναι, κύριε Ιθκάρ, ναι. Ναι, ναι, είχατε ζητήσει και πριν, πράγματι, είναι αλήθεια αλλά όπως είπα Μποστινάρου, Μέγερ, Μπουλάν και βεβαίως θα παραδώσω πάλι την ε, Προεδρία στην Προεδρό μας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε, κύριε Τουργκάη. Συνάδελφοι, πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν αποτελώ τμήμα καμία συνωμοσία και δεν είναι σωστό μερικοί από τους συναδέλφους μας να θεωρούν ότι οι άλλοι είναι συνωμότες. άδικο, δεν είναι σωστό. Δεύτερον, τα καθήκοντά μας είναι όποτε χρειάζεται να οργανώνουμε επισκέψεις ερευνητικές όπως έγινε και έπειτα να γράφουμε εκθέσεις για τα συμπεράσματα των ερευνητικών αυτών αποστολών και μετά να τα εγκρίνουμε. Έχω δει και ο ίδιος και δεν το λέω για να απενευτώ Έχω ζήσει πολλές στιγμές έντασης τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Κοινοβούλιο, αλλά θυμάμαι την περίπτωση της Βουλγαρίας, της Ισπανίας, Πολωνίας και κάθε φορά, ακόμη και αν δεν με βόλευε αυτό, δέχτηκα ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Διότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας. ότι απαιτείται συμβιβασμός. Και αφού πετύχαμε συμβιβασμούς και σε άλλες περιπτώσεις δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην μπορούμε να συμβιβαστούμε και για τη Γαλλικία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή η μόνη δυνατότητα θα ήταν είτε να πούμε δεν θα υπάρξει έκθεση και η υπόθεση της Γαλλικίας δεν θα αναφέρεται καν στην θεσμική μας μνήμη είτε θα εφαρμόσουμε τους κανόνες που έχουμε δεχτεί και στην ερμηνεία της ΑΦΚΟ η έκθεση αυτή θα υποβληθεί από την Πρόεδρο. Αυτοί είναι οι κανόνες και πρέπει να τους εφαρμόσουμε όπως τους έχουν εγκρίνει οι συντονιστές και η Επιτροπή ΑΝΑΦ. Γι' αυτό ζητώ να συμβιβαστούμε και να γίνουν ό,τι αυτά που αποφασίσαμε. Ο κύριος Μέγερ. Σύντομα. Νομίζω ότι πράγματι είναι κυρίαρχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχει τον δικό της βαθμό αυτονομίας και η αντιπροσωπεία. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι τμήμα της διαδικασίας και όταν από τους τρεις οι δύο δεν δέχονται την έκθεση του ενός, γιατί πραγματικά θα γλιτώναμε το χρόνο αν στέλναμε έναν σε κάθε αντιπροσωπεία. Πραγματικά να μην χάνουμε το χρόνο μας. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κάποιοι καταγγέλουμε. Μία αντιπροσωπεία τριών μελών υπάρχει, υπάρχουν δύο οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, επιβάλλεται όμως η άποψη του ενός, της μειοψηφίας δηλαδή. και μετά με τις πλειοψηφίες που θα δημιουργηθούν στις, ε, στις ψηφοφορίες ε, να πω ότι η κυρία Μιράντα ήταν βουλευτής όταν είχε γίνει η έρευνα και ο, ο συνάδελφος που την διαδέχθηκε αναλαμβάνει ακριβώς τις ευθύνες που είχε η προκάτοχός του. Ο κύριος Σαλμπόρ δεν είναι τώρα πια βουλευτής, είναι σαφές, είναι ε, προφανές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει το όνομά του. Ε, αυτός έχει φύγει όμως πολύ καιρό, ενώ η κυρία Μιράντα ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα βουλευτής. Να μην δημιουργούμε μια παράδεκτη κατάσταση. Λοιπόν, ε, το πρόβλημα είναι ότι ε, οι τρεις που πήγαν στην Ισπανία ε, κάνουν μια έκθεση η οποία αντικατοπτρίζει την άποψη μόνον του ενός. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Λο, Κάρλος, για σε και σου νέο en este Parlamento y que estoy aprendiendo, tengo que seguir aprendiendo como tuviste que aprender. Λοιπόν, Πράγματι συγχαίρω τον κύριο Μπολάν για την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει την αυτόματη μετάφραση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για το να μην υπάρχουν οι μεταφράσεις των τροπολογιών επειδή υπάρχει δυνατότητα της χρήσης της αυτόματης μετάφρασης. Τώρα, το πρόβλημα είναι επίσης ότι η Μιράντα ήταν μέλος της Επιτροπής, ενώ Άλμπορ δεν ήταν μέλος της Επιτροπής. Ε, fair play λοιπόν όπως είπε και ο Βίλι Μέγερ. Καλώς. Να διευκρινίσω κάτι γιατί επανερχόμαστε στα θέματα της ε, τροπολογίας της κυρίας Μιράντα. Είναι προφανές ότι οι τροπολογίες που έχουν αποκλειστικά υπογραφεί από κάποιον που δεν είναι πλέον μέλος δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Τροπολογίες οι οποίες έχουν και άλλους συνυπογράφοντες γίνονται δεκτές ε, και βγαίνει το όνομα αυτού που δεν έχει δικαίωμα να έχει το όνομά του εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πλέον διευκρινιστεί. Η τελευταία παρέμβαση από τον ίδιο τον κύριο Μπουλάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν Εύχομαι καλά αρχή καριέρας στο συνάδελφο που μόλις ήρθε, αλλά θέλω να του πω ότι το αυτόματο σύστημα μετάφρασης μας επέτρεψε σήμερα να εκφραστούμε για τις τροπολογίες. Είναι ένα καινούργιο σύστημα, πολύ αποτελεσματικό, αν και όχι τέλειο. Έπειτα, προς τον κύριο Μέγερ ήθελα να πω ότι δεν έχει το μονοπόλιο εδώ μέσα κανείς. Ο καθένας εκφράζεται υπέρ των αναφερόντων. Ο κύριος Μέγερ παρουσιάζει τα πράγματα τμηματικά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ναι μεν υπάρχει αναλογία δύο προς ένα στους ε, μεταξύ αυτών που συμφωνούν και διαφωνούν στην, στην ερευνητική αποστολή αλλά πρέπει να εξισορροπηθούν οι δύο απόψεις. Στο δικό μου κείμενο, όπως και στο κείμενο της Προέδρου, υπάρχει, υπάρχουν και τα δύο, και αυτά που λένε οι αναφέροντες και αυτά που λένε οι υπόλοιποι. Εσείς που μιλάτε για την δημοκρατία όπως και οι άλλοι, πρέπει να ξέρετε ότι από την αρχή έγινε μια ψηφοφορία που δημιούργησε το πρόβλημα. Μια ψηφοφορία που πρέπει και εσείς να τη δεχτείτε, αφού μιλάτε υπέρ της δημοκρατίας και των διαδικασιών που έκρινε την αναφορά αυτή αποδεκτή όχι όμως στα πλαίσια της αποστολής. Με την συνενοχή της γραμματείας τα δύο άλλα μέλη βασίστηκαν σε ένα κείμενο που δεν είχε ακόμη τελειώσει και που ανέφερε τις άτυπες αναφορές που είχαμε αποφασίσει να μην συμπεριλάβουμε. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι τα δύο βασικά σημεία που στα οποία βασίστηκε το πρόβλημα ήταν η συμπερίληψη, η προσπάθεια συμπερίληψη των ατύπων αναφορών που δεν δέχτηκε η αποστολή πριν να φύγει και σε αυτή τη βάση ο πρόεδρος της αποστολής ακόμη και αν είναι μόνος του πρέπει να σεβαστεί την αρχική ψηφοφορία. Αυτό έκανα αρνούμενος στις άτυπες αναφορές και όλες αυτές οι προσπάθειες ακύρωσης και λοιπά των συναδέλφων βασίζονται στο επιχείρημα της συμπερίληψης που ζητάνε των άτυπων αναφορών. Έπειτα. Στην έκθεση που τροπολογούμε και θα ψηφίσουμε υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτών που λένε οι αναφέροντες και αυτών που λένε τα όργανα και εγώ δεν εξυπηρετώ τα συμφέροντα ούτε της τοπικής κυβέρνησης της Γαλλικίας ούτε οποιοδήποτε άλλο. Όπως ο κύριος Μποστινάρου δεν είμαι και εγώ συνομότης κανενός και ό,τι και να μου πείτε εγώ δεν δέχομαι τέτοιες κατηγορίες. Παρακαλώ όχι πάνω από ένα λεπτό κύριε Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ Μπουλόν, γνωρίζω τις μομφές αυτές, τις απορρίπτω τις μομφές κολυσιεργίας. Εσύ έκανες, εσύ προέβησε σε κολυσιεργία, εσύ έλεγες ότι δεν μπορείς να εργαστείς με βάση το αγγλικό κείμενο. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Βέρτμουνα. Να κλείσουμε το θέμα αυτό. Έχει καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα. 16 του μηνός ψηφοφορία των τροπολογιών και του τελικού κειμένου. Περνάω στο σημείο 10, την 1873 του 12, του κυρίου Βέμπερ, Γερμανού πολίτη, για τη χρονομίσθωση εδαφών στην Γαλλία σε Γερμανό γεωργό και για τις διακρίσεις εις βάρος του από πλευράς των τοπικών αρχών ε, λόγω της ηλικία του. Δεν έχει πάρει μέρος στις εργασίες μας ο συγκεκριμένος αναφέρον. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σοτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, δε η κυρία Σοτ. Όντως πρόκειται για θέμα διακρίσεως σε βάση της ηλικίας. Υπενθυμίζω εν συντομία σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να ξεκινήσει η προσφυγή για παραβίαση διατάξεως της συνθήκης όταν δεν εφαρμόζονται ή μάλλον δεν έχουν περάσει το εθνικό δίκαιο σωστά η, εθνική, η, ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόκειται για την οδηγία 78 του 2000. Εξετάσαμε την μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο στη Γαλλία για την επιμέρους η υπόθεση πρόκειται για τον Γαλλικό Αγροτικό Κώδικα που προβλέπει ότι για την μίσθωση γεών προβλέπει ότι οι αρχές μπορούν να εξετάσουν και την ηλικία. Η ίδια η Γαλλική Αρχή, η αρμόδια Γαλλική Αρχή κρίνει που λέει ότι έχει εφαρμοστεί η βασική νομοθεσία κατά των διακρίσεων στη βάση ηλικία. Και αν κάποιος θεωρήσει ότι αδικείται λόγω ηλικία, αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται καλά ο γαλλικός νόμος. Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρόκειται για εφαρμογή σε μεμονωμένη περίπτωση που υπάγεται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και ενδεχομένω των εθνικών δικαστηρίων. Ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε μεμονωμένη περίπτωση και να δούμε εάν ο νόμος εφαρμόστηκε σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ωστόσο μια ερώτηση. Αυτό το όριο ηλικίας ισχύει μοναχά για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και για Γάλλους πολίτες. Γιατί, συγγνώμη, μια στιγμή, παρακαλώ, άμα θέλετε να κάνετε πηγαδάκια, εξέλθετε της αιθούσεις. Έχουμε συνάδελφο που ομιλεί. Δείξτε σεβασμό στο πρόσωπο των παρεμβενόντων. Συνεχίζει ο κύριος Γιάρ. Βεβαίως υπάρχει οδηγία κατά των διακρίσεων που ορθώς εφαρμόζεται από τη Γαλλική Δημοκρατία, ένας τώρα που είναι 61 ετών, 61, και θέλει να μισθώσει η αγροτική γη, του λένε «Α, είσαι πολύ μεγάλος η ηλικία». Αναρωτιέμαι, τέλος πάντων, τι νόημα έχει τότε η οδηγία κατά των διακρίσεων στη βάση της ηλικίας. Δεν θεωρώ άλλωστε ότι είναι μεμονωμένη υπόθεση γιατί έχουμε λάβει πολλές σχετικές αναφορές. Και τελικά πού αρχίζει να είναι κανείς ηλικιωμένος. 61 ετών. Στη Γερμανία η ηλικία ταξιοδότηση είναι 67 ετών. Και πώς θα απαγορεύσει κάποιον να εργάζεται λόγω ηλικίας. Και άλλωστε εδώ πρόκειται και για την ελευθερία του επιχειρήν. Η απάντηση αυτή μου φαίνεται υπερβολικά ελαφριά της ε, Επιτροπής και λέει ότι είναι μεμονωμένη περίπτωση. Αλλά δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη περίπτωση, διότι γενικά στην εκμίσθωση αγροτικών γιών λαμβάνεται υπόψη το όριο ηλικία. Για μένα αυτό είναι μορφή διακρίσεως. Αν μάλιστα τώρα πρόκειται για καρτέλ ή πρόκειται για παραβίαση της αρχής εγκαταστάσεως, είναι και αυτό μια υπόθεση που πρέπει να εξεταστεί. Πώς μπορείς να απαγορεύσει κάποιον να ασκήσει το επάγγελμα του αγρότη. Τουλάχιστον λοιπόν να διατηρηθεί ανοιχτή και ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό ποιες συνθήκες, υπό ποιους όρους θα παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ προφανώς η πρακτική εφαρμογή, στην πράξη εφαρμογή δηλαδή, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που έχει αποφασίσει και η ίδια η Γαλλική Δημοκρατία δηλαδή την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τέλο πάντων η απάντηση αυτή δεν μου αρκεί. Να μην σας πω ότι μου σηκώνονται οι τρίχε μόλις την ακούω. Και εγώ είμαι σχεδόν 61 και θα, θα μου πούνε τώρα όχι απαγόρευση επαγγέλματο. Εσείς, Βίκτορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απάντηση της Κομισιόν είναι λίγο περίεργη. Πρώτον, είτε υπάρχει παραβίαση είτε δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι πρόκειται για παραβίαση της οδηγίας όταν φτάσει μια κρίσιμη μάζα αριθμού παραβιάσεων, αλλιώς όμως δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Πώς το ερμηνεύεται δηλαδή. Αν θεωρείτε ότι ένα κράτος μέλος, διότι γενικά τώρα το 2014 η Ρουμανία θα ανοίξει την αγορά της στους ενωσιακούς πολίτες. Αν θεωρήσετε ότι μπορεί ίσως η Ρουμανία να παραβιάσει τον νόμο όταν φτάσουμε στις 10, 100, 1000 περιπτώσεις μόνο θα θεωρείτε ότι παραβιάζεται ο νόμος. Δεν έχει σημασία ο αριθμός για να κρίνουμε αν υπάρχει παρανομία ή όχι. Αυτό μου φαίνεται προφανές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ περιγραφής και εφαρμογής. Ένα είναι να λέμε πολύ σωστά εφαρμόζει η Γαλλία την οδηγία για την ίση μεταχείριση με, ή άνηση μεταχείριση με βάση την ηλικία και άλλο να λέτε μα είναι μόνο μια περίπτωση και δεν έχει σημασία. Όχι, σε δικαστήριο. Για το δικαστήριο είτε υπάρχει παρανομία είτε δεν υπάρχει. Και μετά λαμβάνεται η απόφαση. Η εφαρμογή δεν συνίσταται στο να λέμε ότι κάποτε ίσως θα εφαρμοστεί σωστά. Αφοροβλέπονται εξαιρέσεις δηλαδή. Εξαιρέσεις σημαίνει παραβίαση του νόμου. Εγώ δεν είμαι μεν δικηγόρος αλλά και για κάποιον που δεν έχει πολλές νομικές γνώσεις καταλαβαίνουμε ότι και μία μόνο παρανομία αρκεί για καταδίκη. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Μήπως η Κομισιόν θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να λάβω πάλι το λόγο. Επιθυμώ να περάσω ίσως σε περισσότερες λεπτομέρειες για να κατανοήσετε καλύτερα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφενός, δεν πρόκειται όντως για το ερώτημα αν είναι μία υπόθεση, δύο ή χίλιες. Το ερώτημα είναι κατά βάση μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διοίκηση των κρατών μελών. Όχι, δεν μπορεί. Η Κομισιόν μπορεί να επιτιμήσει την χώρα μέλος ή την κυβέρνηση αν δεν εφαρμόζει σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πολύ πιο δύσκολο θα το ερώτημα που όμως δεν αντιμετωπίζει σχεδόν ποτέ η Κομισιόν με ελαχίστες εξαιρέσεις εφόσον πρόκειται για διαδικασία επί παραβιάση των συνθήκων. Αν υπάρχουν για παράδειγμα πολλές εσφαλμένες αποφάσεις. Δεν παρεμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δει ότι υπάρχουν 10 ή και 100 υποθέσεις όπου ο νόμος ερμηνεύεται με τρόπο όπου η Κομισιόν θεωρεί ότι ε, δεν ανταποκρίνεται στην αρχική έννοια της οδηγίας. Πρέπει πρώτα να τα κάνουν τα πράγματα αυτά οι εθνικές αρχές. Αυτό βεβαίως γενικά. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση να σας εξηγήσω την οδηγία. Η οδηγία επιτρέπει στις χώρες μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς στην βάση της ηλικία. Αυτό ίσως να μην έχει καταστεί απόλυτα σαφές, αλλά το είπε στην απάντησή της η Κομισιόν. Η οδηγία λέει καθαρά ότι μπορεί η ηλικία να είναι λόγος διακρίσεως. Βεβαίως όλοι έχουμε κάποια ηλικία. Επομένως όλοι μπορούμε κάποια στιγμή να πέσουμε θύματα της διακρίσεως. Αυτό σημαίνει ότι για την ηλικία πρέπει αυτή να υπακούει και σε συγκεκριμένα κριτήρια. Πότε δηλαδή αποτελεί λόγο διακρίσεως και πότε αποτελεί απλώς κάποια εξειδίκευση. Επ' αυτού η οδηγία λέει ότι σε ορισμένου τομεί, άλλωστε πρόκειται μοναχά για εργασία και απασχόληση, εκτό εργασία και απασχόληση δεν υπάρχει καμία προστασία κατά τη διακρίσεω σε βάση τη ηλικία. Για την απασχόληση υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, η οδηγία επιτρέπει στον τομέα της πρόσβασης στην απασχόληση, για παράδειγμα για κάποια εκπαίδευση ή να υπάρχουν κάποια ανώτατα, κάποια ανώτατα όρια πρόσβασης σε ένα επάγγελμα. Αυτά καταρχήν επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια της χώρας μέλους και αυτήν τη διακριτική ευχέρεια την έχει περιλάβει στον αγροτικό της κώδικα η Γαλλία ώστε να επιβάλλει κάποια όρια σε αυτή την δραστηριότητα της ε, καλλιέργειας αγροτικών εδαφών. Εάν ο πολίτης δεν συμφωνεί, μπορεί να στραφεί στις αρχές και ή στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν πρώτα ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο και μετά το Εθνικό Δικαστήριο μπορεί να υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως είπα όμως η Κομισιόν εξέτασε, ερεύνησε το θέμα και διαπιστώνει ότι η Γαλλική Δημοκρατία έχει την ελευθερία να επιβάλλει κάποια όρια ηλικία στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν, επαναλαμβάνω, η χώρα μέλο διαθέτει ορισμένε ελευθερίε. Αυτό άλλωστε είναι και το περιεχόμενο τη οδηγία, ότι δεν επιβάλλει τα πάντα, αλλά ότι αφήνει ευχέρειε, αφήνει διακριτική ευχέρεια στι χώρε μέλη. Και ο Βίκτορ και ο Πέτεριά ζητούν ξανά το λόγο. Αλλά σύντομα. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Σήμερα θα γράψω επιστολή στη ρουμανική κυβέρνηση που θα λέει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2014 πρέπει η Ρουμανία να ακολουθήσει τον γαλλικό δρόμο. Αν είναι τόσο χαλαρή η ερμηνεία, γιατί να μην κάνει και η Γερμανία το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανοιχτή σας ερμηνεία ήξερα και από παλιά ότι ντούρα λέξ σεντ Αν αυτό δεν ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εντάξει, εφαρμόστε το γαλλικό πρότυπο. Πέτερ Γιάρ. Εγώ παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα εξετάσω και περί τι άλλος πρόκειται. Δεν πρόκειται ούτε για συντροξιοδότηση, ούτε για παροχές υπηρεσιών μια χώρας, αλλά ότι κάποιο έχει ε, ε, στην ε, κυριότητά του έδαφος, θέλει να το μισθώσει το έδαφος αυτό, το ακίνητο αυτό σε κάποιον άλλο και το κράτος έρχεται και λέει όχι αυτός ο άλλος είναι πολύ δικαιωμένο. Πρόκειται όμως για σχέση ιδιωτικού δικαίου. Και πού θα βάλουν το όριο. 30, 40, 50. Βεβαίως κάποια ηλικία έχουμε όλοι. Εφόσον ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο, τότε μου φαίνεται ότι είναι εντελώ περιττή πλέον η οδηγία περί μη διακρίσεων. Να παραμείνει ανοιχτή λοιπόν. Πρόκειται καθαρά για ιδιωτική σχέση μεταξύ δύο ιδιωτών. Και ξαφνικά κατέβεται το κράτο και λέει: Όχι, εσύ, ένα από του δυο δηλαδή, είναι υπερβολικά ηλικιωμένο. Αυτό σημαίνει όμω παρέμβαση στην ε, ιδιοκτησία μου, παρέμβαση στην ε, επαγγελματική μου δραστηριότητα και ούτω καθεξής. Πραγματικά λέω ότι μου σηκώνονται τρίχες όταν τα πω αυτά τα πράγματα. Και καλά το είπε ο Μποστινάρου, ότι άμα είναι έτσι τότε καλά θα κάνουν και όταν έρθουν οι Βούλγαροι ή οι Ρουμάνοι εργάτες να δουλέψουν στη Γερμανία, τότε να βγάλει και η Γερμανία ένα φετφά που να λέει άμα είναι πάνω από 22 χρόνια δεν μπορούν να δουλέψουν. Μάλιστα, Παραμένει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά. Α, Πέτερ, άκουσέ με. Και σε σχέση με αυτά που είπες εσύ και με αυτά τα οποία είπε ο Πίτερ, θα αφήσουμε ανοιχτή λοιπόν τη συγκεκριμένη αναφορά. και να ζητήσουμε να στείλουμε μία αναφορά ε, για περαιτέρω πληροφόρηση από τις γαλλικές αρχές. Καλώς ήρθατε κυρία Παλιαδέλη. Οι επτά εξ ονόματος των καθηγητών βιοχημίας για την παράταση του κανονισμού για την δροσόφυλλο των φρούτων και για τα, τους κτηνιατρικούς ελέγχους του συγκεκριμένου είδους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο στην αναφέρουσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κάποιες εξηγήσει. Να σας εξηγήσω την σημασία της ε, προκειμένης αναφοράς. Η έρευνα με βάση την ε, ντροσόφυλλα μελαγκάστερ είναι ουσιοδέστατη και απαραίτητη για την ιατρική έρευνα. Γιατί χρησιμοποιείται η δροσόφυλλα του τύπου μελανογκάστερ. Η γενετική σύνθεση ή αν θέλετε η δόμηση των, ε, του γονιδιώματος της δροσόφυλλα μελανογκάστερ είναι πολύ παρόμοια με το ανθρώπινο γονιδίωμα. Σε πολλά σημεία λοιπόν είναι πολύ συγκρίσιμη. Επίσης, η μελανογκάστερ έχει πολύ σύντομη διαδοχή, γενεών, δηλαδή έχει πολύ σύντομη διάρκεια ζωής και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερευνητές. Η έρευνα με την τροσόφυλλα μελανογκάστερ, δηλαδή η ιατρική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει τις χέρειες λόγω των συνοριακών κτηνιατρικών ελέγχων επηρεάζεται πολύ σημαντικά για να μην πω ότι παρεμποδίζεται και καμιά φορά ματαιώνεται εντελώς. Το ερώτημα είναι γιατί η οδηγία 491 έχει εισαχθεί κατά τη γνώμη μας για την προστασία των καταναλωτών έναντι ενδεχόμενων κινδύνων. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να επηρεάσει η δροσόφυλλα τους καταναλωτές. Για την προστασία καταναλωτού δεν έχει απολύτως καμία σχέση η ε, μιγούλα αυτή των φρούτων. Το άλλο ερώτημα είναι τι μπορούν να εξετάσουν οι κτηνίατροι. Τίποτα. Αυτές οι φυλές των μηγών παράγονται στα εργαστήρια υπό συνθήκες στηρότητας και αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια όπου πάλι το περιβάλλον είναι απόλυτα αποστηρωμένο. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα, από τότε που άρχισαν μάλλον οι κτηνιατρικοί έλεγχοι το 2009, έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικότατες παρεμβάσεις, υπερβολικά μακρά η διάρκεια των μεταφορών, οι φυλές των εντόμων φτάνουν με πολύ μεγάλες ζημιές, είτε απολύτως κατεστραμμένες ή πάντως σχεδόν άχρηστες πλέον για την έρευνα. Επομένως δεν μπορούν οι ερευνητές πλέον να τις χρησιμοποιήσουν για ε, ερευνητικούς σκοπούς. Ουδής μπορεί να κρίνει βεβαίως τι ακριβώς συμβαίνει. Οι διάφοροι μεταφορείς, είτε πρόκειται για την FedEx ή την UPS ή τα διεθνή ταχυδρομεία ή το DHL λένε ότι δεν μπορούμε πλέον να παραδίδουμε εντός των χρονικών προθεσμιών που μας ζητάτε διότι γίνονται οι συνοριακοί ε, κτηνιατρικοί έλεγχοι. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορούν να εξετάσουν οι κτηνίατροι, τι θα εξετάσουν σε αυτά τα απειροελάχιστα έντομα. Και όπως είπα, οι καταναλωτές δεν έχονται σε καμία απολύτως επαφή με τα έντομα αυτά. Γι' αυτό και υποβάλλουμε την αναφορά αυτή με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να πάψουν αυτές οι δυσκολίες που τόσο πολύ εμποδίζουν την έρευνα και ότι οι μύγες της, ε, του τύπου δροσόφυλλα μελανογκάστερ που διακινούνται και διαμεθοριακά θα μπορέσουν επιτέλους να εξαιρεθούν από τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Από την Κομισιόν. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας όλοι. Βεβαίως κατανοούμε τις ανησυχίες της αναφέρουσης. Τη μελετήσαμε την αναφορά πολύ προσεκτικά και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προτεραιότητα και δική μας είναι να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στις ζωικές μεταφορές για να μην υπάρχουν πρόσθετα βάρη των μεταφορέων είτε πρόκειται για μεγάλα ζώα είτε για έντομα όπως δροσόφυλλα μελανογκάστερ που λένε. Παρόλα αυτά η νομοθεσία καθορίστηκε το 1991 και η οδηγία 9146 προβλέπει τον κτηνιατρικό έλεγχο όλων των ζών των ζώων στα σύνορα διότι θεωρείται μεγάλος κίνδυνος η μεταφορά τους για τη διάδοση ασθενειών. Τώρα αναθεωρούμε, επανεξετάζουμε τους ελέγχους αυτούς, η νομοθεσία για τους ελέγχους στα σύνορα και έχουμε προβλέψει σε μία πρόταση που σε λίγο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τη δυνατότητα εξαιρέσεων από τους κτηνιατρικούς ελέγχους για συγκεκριμένα είδη που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αν η εξαίρεση αυτή εγκριθεί από όλους ή όχι. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι δεν εισάγονται μόνο έντομα για επιστημονικούς λόγους, εισάγονται έντομα και για ανθρώπινη κατανάλωση και γι' αυτό Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας αν έντομα, έστω και αν παράγονται από εργαστήρια, μπορεί να καταναλωθούν από ανθρώπους. Θα το δούμε αυτό όμως στο μέλλον, όταν θα γραφτούν οι συγκεκριμένες διατάξεις που αναθεωρούμε. Προς το παρόν το σκεφτόμαστε, το εξετάζουμε και θα παρακολουθήσουμε τις εισαγωγές εντόμων για να δούμε αν υπάρχει όντως κάποιος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή όχι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μου αρκεί τόσο πολύ αυτή η απάντηση εξετάζοντας αυτόν τον θεωρητικό κίνδυνο ότι ενδεχομένως κάποια έντομα μπορεί να ξεφύγουν από ε, τα πειραματικά εργαστήρια και να φτάσουν στην ανθρώπινη κατανάλωση, μα σε κάθε κουτί με μπανάνες έχει έντομα μέσα. Εγώ νομίζω ότι εκεί η έλεγχη είναι πολύ λιγότερο καλή από ό,τι εδώ, από ό,τι στην προκείμενη περίπτωση. Οι εκπρόσωπος των αναφερόντων και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και βραβευμένοι με βραβεία Νόμπελ στην βάση πειραμάτων με τα έντομα αυτά έχουν κάνει σοβαρότατες έρευνες, έχουν πάρει ενδεχομένω και το βραβείο Νόμπελ για αυτές και επομένως τα έντομα αυτά αποτελούν ένα είδος, πώς να πω, τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής έρευνας. Και η Ευρώπη ως έδρα επιστημόνων υφίσταται ζημιά, εφόσον δεν το προσέξουμε αυτό. Πρόκειται για ένα έντομο, στα γερμανικά μάλιστα λέγεται Eintagsfliege, η μήγα της μιας ημέρας. Έχει τόσο σύντομη ζωή, οι γενναίες διαδέχονται μια την άλλη ταχύτατα, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την έρευνα. Έχει πολύ λίγο χρόνο λοιπόν η μίγα αυτή για να διέλθει τα σύνορα. Τα πανεπιστήμια που διαλέγονται μεταξύ τους ενδιαφέρονται και για τις συγκεκριμένες ειδικέ φυλές των μυγών αυτών, από αυτές παράγουν έντομα, εάν κάποιο πανεπιστήμιο κάπου στον κόσμο έχει, θέλει μάλλον να χρησιμοποιήσει ένα έντομο, μια τέτοια μύγα η οποία έχει 5, 6, 7 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα το ζητήσει να το βρει και να το λάβει από κάπου αλλού στον κόσμο, που μπορεί να μην το έχει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το ζήτημα είναι εάν τα έντομα αυτά φτάσουν είτε με βλάβες είτε και νεκρά, δεν έχει απολύτως πλέον καμία αξία για το εργαστήριο. Και πάει περίπατο, όπως εξήγησε και η αναφέρουσα ολόκληρη έρευνα. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια εναρμονισμένη αντιμετώπιση στα σύνορα. Σε ορισμένα σύνορα τα πράγματα πάνε καλύτερα, σε άλλα πάνε χειρότερα. Και από αυτή την έννοια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό λοιπόν αυτό. Επίσης είναι πολύ διαφορετικά τα τέλη. Τα πανεπιστήμια εξυπηρετούν το ένα το άλλο χωρίς κόστος, δωρεάν. Όμως σε ορισμένα αεροδρόμια ζητείται η καταβολή υπέρογκων τελών για να διέλθουν τα έντομα. Αναμένοντα εν πάση περιπτώσει την αναθεώρηση αυτή τη οδηγία, δεν θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στι χώρε μέλη ώστε η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων να γίνει με τρόπο όμοιο εναρμονισμένα να εξυπηρετηθεί το δίκτυο αυτό των επιστημόνων, να βελτιωθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και από το Ενωμένο Βασίλειο υπάρχουν εδώ ευρωβουλευτές οι οποίοι παρακολουθούν την αναφορά αυτή με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει και εκεί πάρα πολύ σημαντική ανάγκη από τα έντομα αυτά. Φοβούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ιδιαίτερα παθητικό ρόλο και παίζει το ρόλο του θεατή μέχρι ότου δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχουν και κατευθυντήρες γραμμές, μπορούν να εκδώσουν λοιπόν κατευθυντήρες γραμμές, guidelines, που να εξηγεί στι χώρε μέλη ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικές ώστε όσοι θέλουν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αυτές και να απλοποιηθούν, τουλάχιστον να μην κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν με ικανοποιεί λοιπόν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν με ικανοποιεί και η πρακτική εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε υποβάλει το θέμα αυτό στην Επιτροπή Γεωργίας εδώ και καιρό. Η Επιτροπή Γεωργίας είπε δεν κάνουμε τίποτα μέχρι ότου υπάρξει αναθεώρηση της οδηγίας. Αυτό όμως εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν είναι θέση αυτή η Επιτροπή Γεωργία. Θα μπορούσε η Επιτροπή Γεωργία να πει μάλιστα και εμεί θέλουμε να προχωρήσει. Ε, σχεδόν ένα χρόνο έχουμε παραλύσει εδώ διότι η Επιτροπή Γεωργίας αρνήθηκε να αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό το πράγμα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. για την επισήμανση ό,τι αφορά την Επιτροπή για την Αγροτική Ανάπτυξη. Κύριε Ποστινάρου. Thank Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ακούγοντας την απάντηση της Κομισιόν, σκέφτηκα να απαντήσω στα ρουμανικά, διότι θα αναφέρω μερικές λεπτομέρειες ανεκδοτολογικές. Όλοι έχουν καλές προθέσεις, αλλά εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Στη Ρουμανία, στη Ρουμανία λέγω, υδροσόφυλλα, ονομάζεται μεθυσμένη μίγα, διότι περιφέρεται εκεί όπου στα Ινοπία Πώς μπορεί κανείς να εμποδίσει τη δροσόφυλλα να περάσει σύνορα. Συνήθως οι δροσόφυλλες δεν μπορούν να... Ε, τώρα μας λένε ότι οι δροσόφυλλες δεν μπορούν να περνάνε τα σύνορα χωρίς άδεια. Πώς τότε τις επιτρέπετε να κυκλοφορεί σε τόσο μεγάλους αριθμούς γύρω από τα Ινωπία το ελέγχει και αυτό η Κομισιόν. Χρειάζονται πιστοποιητικά. Εδώ γίνεται προσπάθεια νομοθετικής διευθέτησης και των παραμικροτέρων λεπτομεριών και αυτό καταλήγει γελίο τελικά. Η Κομισιόν δίνει ιδιαίτερη σημασία φαίνεται και προσοχή στη δροσόφυλλα μελανογκάστερ αλλά Υπάρχουν και οδηγίες για τον ανταγωνισμό, για το περιβάλλον, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι οποίες δεν γίνονται σεβαστές, όπως ακούσαμε από άλλες αναφορές σήμερα. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίος γιατί πολλές φορές έχει δίκιο η Ένωση αλλά η γραφειοκρατία των Βρυξελών μερικές φορές δυσκολεύει τα πράγματα χωρίς λόγο για τους ερευνητές παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ιδιαίτερο παράδειγμα αυτό που συζητάμε σήμερα. είναι ένα θέμα που έχει πολύ μικρή σημασία και πολύ λίγες εδώ μηδαμινές υγειονομικές επιπτώσεις και ζητιέται τέτοια διευθέτηση. Εδώ είναι θέμα κοινή λογικής. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν ανακατεύεται με τέτοια θέματα. Πρέπει να δεχτεί και η Κομισιόν ότι οι επιστημονικές έρευνες όπως λέει και η αναφέρουσα ή αναφερόμενη δικαιολογούν την εξαίρεση. Δεν χρειάζεται άλλη εξέταση. Πρέπει να αφήσουμε τους ερευνητές να χρησιμοποιούν την δροσόφυλλα μελανογκάστερ και να μην τις φέρονται σαν να είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, κυρία Γκρός, θέλετε να πείτε κάτι. Sehr gerne möchte ich äh, äh, zu den Ausführungen der äh, der Vertreterin Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ουσία αυτό το οποίο είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να επαληθευτεί το αν συνιστούν συγκεκριμένο κίνδυνο ή ε, τα συγκεκριμένα αυτά έντομα. Ε, φοβάμαι ότι δεν έχει ενημερωθεί σωστά η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Εκτρέφονται, να το πω έτσι, τα, τα, τα έντομα αυτά κάτω από ειδικέ συνθήκες ασυπτικές και ε, ε, αποστέλλονται σε αντίστοιχα εργαστήρια και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος γύρω από αυτό. Και έχει αποδειχθεί ότι οι μύγες αυτές δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα και κανένα κίνδυνο. Και παρόλα αυτά το 2009 ξεκίνησε ο τελωνιακός έλεγχος, ο μεθοριακός έλεγχος και ιδίω κτηνιατρικός έλεγχο, τι δουλειά έχουν οι κτηνίατροι να ελέγχουν τις μύγε δροσόφυλλα στα αεροδρόμια. Δεν μπορώ να κατανοήσω και κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει. Το γεγονό είναι πάντως ότι υφίσταται τι αρνητικέ συνέπειες η έρευνα, διότι δεν μπορούν τώρα πλέον άνευ εταίρου να ανταλλάσσουν ε, αποστολές τέτοιων μυγών και επομένως τίθεται σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή έρευνα. Επανέρχομαι στα όσα είπε ο βουλευτής κύριος Βίλαντ. Μα θα πρέπει να ελεγχθεί και το κάθε πουλόβερ, διότι μπορούν να μπουν μέσα και να κρυφτούν αυγά μυρμηγκιών που προέρχονται από άλλες ε, χώρες και μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ πιο επικίνδυνα έντομα τα οποία κρύβονται για παράδειγμα στα ρούχα των ε, περιηγητών, των τουριστών που επανέρχονται από μακρινά εξωτικά ταξίδια και όχι από έντομα τα οποία έχουν καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί μέσα σε απόλυτα αποστηρωμένες συνθήκες. Επαναλαμβάνω ότι η έρευνα στην Ένωση επηρεάζεται αρνητικά και στο κάτω της γραφής όλοι οι πολίτες έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον να ε, προωθηθεί η έρευνα η οποία μπορεί να διευκολύνει και την ε, ε, θεραπεία ασθενειών όπως το Alzheimer ή ο καρκίνος. We have to deal with... Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταχύτερα το θέμα. Σωστό αυτό. Δέχομαι λοιπόν την πρόταση του γραμματέα μας εδώ να απευθυνθούμε στον Επίτροπο που ασχολείται με το θέμα, διαβιβάζοντας μαζί και την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και να του ζητήσουμε να πράξει πάντο δυνατό, όχι να παραμένει απαραίτητα την οδηγία η οποία θα εκπονηθεί τους επόμενους μήνες ή τέλος πάντων. Να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα το δυνατόν ταχύτερο, διότι ε, εμείς ε, σεβόμαστε βαθύτατα την επιστημονική έρευνα. Ας προχωρήσουμε στην υπαριθμόν 8. που είναι ισπανική αναφορά με παρόμοιο αντικείμενο που είναι ο αναφέρον σας παρακαλώ να μπορείτε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Λάβαμε υπόψη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τέλος του Αυγούστου του 2013 και γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε αποστείλει αρκετά σε επιστολές στην Γραμματεία και της Επιτροπής σας, μεταξύ των οποίων και την άποψη της Επιτροπής Προβλέψεων της, ε, του συγκεκριμένου τομέα των εσπεριδοειδών, όπως επίσης και τις απόψεις της ΕΨΑ ε, για την ασθένεια αυτή των εσπεριδοειδών που λέγεται black spot, γκινιάρδια σιτρίκαρπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη παρουσιάσει μια πρόταση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, δημιουργία ε, ενός συγκεκριμένου ταμείου για την καταπολέμηση τέτοιου είδους ε, απειλών και ήδη από τις 14 Δεκεμβρίου του 2000 11 είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες και τέθηκε επίσης και το θέμα του ιδιοκτήτη, αν θέλετε, της, του κατόχου της συγκεκριμένης ε, ε, ενεργούς ουσίας και ε, από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν εξελίχθησαν σωστά. Εμείς έχουμε προβλήματα στην Βαλένθια όπως και στην υπόλοιπη Ισπανία. Δεν έχουμε αρκετές ενεργές ουσίες αδειοδοτημένες για την καταπολέμηση των ασθενειών των δέντρων, των φυτών. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή και κάθε χρόνο η κυβέρνησή μας πρέπει να εκδίδει εξαιρετικές άδειες αποκλήσεως από την κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη συμβαίνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ε, με την εμπορία των συγκεκριμένων ουσιών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αντιμετώπιση νέων ασθενειών που προέρχονται από τρίτες χώρες ε, και είναι συνέπεια των εισαγωγών των φυτικών προϊόντων τους και μετά και από την απόφαση σχετικά με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα προστασίας των φυτών από ασθένειες βελτιώνεται η προηγούμενη απόφαση του 2009 αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται πλήρως σαν παράδειγμα δεν ε, λαμβάνονται υπόψη όλα τα τεχνικά επιχειρήματα και υπάρχουν άλλα επιχειρήματα τα οποία ε, λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ίσχυε και στην Οδηγία 2029. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη δημοκρατία της, Νοτιού Αφρικής ε, για, την... για την εισαγωγή εσπεριδοειδών που έχουν θυγεί από την Κιγνάρδια Σιτρίκαρπα Ήδη η Επιτροπή είχε, πάρει, είχε ανακοινώσει ότι θα πάρει μέτρα σε σχέση με την εισαγωγή εσπεριδοειδών που υποφέρουν από το λεγόμενο black spot. Σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυξάνεται ο αριθμός του εντοπισμού μετά από το σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των εσπεριδοειδών που έχουν φυγεί από τη συγκεκριμένη ασθένεια ό,τι φαίνεται όμως η Νότια Αφρική συστηματικά αγνοεί τα αιτήματα βελτίωσης και αντιμετώπισης του προβλήματος από πλευράς των Βρυξελών. Ε, και δεν έλαβε κανένα μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως η κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγών. Η, Αμερικανική, η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση δεν παρέχει πλέον εγγυήσεις ασφάλειας αλλά μετά την πέμπτη ε, φορά που εντοπίστηκε η ασθένεια αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε εκ νέου την κατάσταση, δεν πήρε όμως κανένα μέτρο. Είπε ότι από πλευράς ε, της ε, Νοτιού Αφρικής η απόφαση εξαγωγής προϊόντων από περιοχές αποκλειστικά προστατευμένες από τη συγκεκριμένη ασθένεια έδειξε ότι την ικανοποιούν. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση έχει χειροτερεύσει και ήδη από τον μήνα Οκτώβριο έχουμε 34 εντοπισμούς φρούτων τα οποία έχουν φυγεί από τη συγκεκριμένη αυτή ασθένεια. Και στις 20 Νοεμβρίου υπήρξε μια απαράδεκτη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με την εισαγωγή των ε, προϊόντων εσπεριδοειδών και βλέπουμε ότι έχουν εξαχθεί μέσα σε ένα μήνα 150.000 τόνοι και ε, προβλέπεται μέχρι το τέλος του χρόνου άλλες 200.000. Συνεχίζεται η απαράδεκτη τακτική δηλαδή της Νοτιού Αφρικής και απλά έχουν απαγορευτεί κάποιες πολύ μικρές ποσότητες δηλαδή το 1,36 της χιλής του συνόλου των εξαγωγών της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, είναι μια κοροϊδία εις βάρος της ευρωπαϊκής ε, ε, φυτοπαραγωγής. Εμείς δεν απειλούμε, ε, απλά θεωρούμε ότι μας έχει προδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει πάρει μη επιστημονικές αποφάσεις αντίθετες με τις αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής για την υγιεινή των τροφίμων και ε, με τεράστιες συνέπειες για την ε, παραγωγή ε, στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιο τρόπο να παραμείνουν σε λειτουργία οι δυνατότητες παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των εσπεριδοειδών απαιτείται να αναλυφθούν οι ευθύνες ε, ε, που αναλογούν στους αρμόδιους επιτρόπους και όχι ε, θα έλεγα γιατί όχι και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει έκτακτα μέτρα και από άλλες τρίτες χώρες για τη συγκεκριμένη ασθένεια όπως την Αργεντινή ε, αυτό σημαίνει κόστος για την διασφάλιση των εξαγωγών της, ενώ αντίθετα στην Νότια Αφρική επιτρέπονται τα πάντα. Και τέλος υπάρχει και η ακατανόητη ε, άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου ε, για τις θυγμένες περιοχές επιτόπου, κάτι το οποίο δεν θα κοστίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ακριβώς συμβαίνει με άλλες μεγάλες γεωργικές δυνάμεις, κάτι το οποίο διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ε, την ίδια την χώρα εξαγωγής. Και ζητάμε επίσης και την κατάργηση του μηχανισμού ανοχής ε, στις ε, εισαγωγές και με την εφαρμογή αυτού του μέτρου δυστυχώς υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των, Ευρωπαίων παραγωγών στον τομέα και των εσπεριδοειδών και γενικότερα της παραγωγής φυτικών προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν με με μεγαλύτερη αυστηρότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και ε, να υπάρξει και αμοιβαιότητα σε σχέση με, την, με το σύστημα, να επιτραπεί λοιπόν το σύστημα αδειοδότησης έκτακτα συγκεκριμένων ουσιών σύμφωνα και με τις αποφάσεις της ΦΑΟ και φυσικά σεβόμενοι τους διεθνείς κανονισμούς για την κυκλοφορία φυτοπροστατευτικών ουσιών ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ο κύριος... Η Αρένα να πάρει λόγο να, μας εξηγήσει. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Θέσατε σημαντικά θέματα σε δύο διαφορετικούς τομείς τους οποίους διέπουν διαφορετικές νομοθεσίες. Το πρώτο που θέσατε ήταν για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την διαθεσιμότητα των ενεργών ουσιών, καθώς και την δυσανεξία σε ό,τι αφορά ορισμένους από τους παράγοντες αυτούς. Μιλήσατε επίσης και για ένα θέμα ε, υγείας των φυτών. Για αυτό όμως θα δώσω τον λόγο στον συναδελφό μου. Πολύ σωστή χρονική στιγμή για την παρέμβασή σας. όσον αφορά έκτακτες χρήσεις. Ήδη η βουλευτής Πάολα Δικάστρο έκανε σχετικό σεμινάριο για τις χρήσεις αυτές. Και εκεί η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η έκθεση, η οποία δυστυχώς έχει καθυστερήσει και δεν το αρνούμεθα αυτό, θα εγκριθεί και θα δημοσιευτεί τον Γενάρη. Ωστόσο, ήδη μπορούμε να πούμε ότι στην έκθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο να δίνει επιχορηγήσεις για τις ελάσσονες αυτές χρήσεις, για τον συντονισμό μεταξύ των χωρών ε, μελών και με ένα πρώτο ποσό 400.000 ευρώ τον, ευρώ τον μήνα. Αυτό λοιπόν θα επιτρέψει την αύξηση της εναρμόνισης και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών και ενδιαφερομένων μερών για να διευκολυνθεί ακριβώς αυτή η υπόθεση των ε, ελασσόνων χρήσεων. Ωστόσο, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει έργα έρευνας και συντονισμού που λέγονται Eranet για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών και αυτή η προσπάθεια θα αρχίσει πάλι από τον επόμενο Γενάρη, θα, θα διαρκέσει τρία χρόνια και με δύο εκατομμύρια προϋπολογισμό. Άρα ξεκινούν και προχωρούν διάφορες δραστηριότητες για τις ε, ελάσσονες χρήσεις και είμαστε πεπισμένες ότι καλύτερος συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών ε, θα επιτρέψουν ήδη να επιτύχουμε πολλά. Διότι το βασικό θέμα είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά οι χώρες μέλη δεν αναγνωρίζουν τις εγκρίσεις που έχουν ε, χορηγήσει λόγω έλλειψης πληροφοριών και έλλειψης συντονισμού. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι στην Ευρώπη έχουμε παραπάνω από 400 ενεργές ουσίες που έχουν εγκριθεί. Έχει βελτιωθεί λοιπόν πολύ η κατάσταση από το 2010 περίπου, όταν εσείς καταθέσατε την αναφορά σας. Έκτοτε έχουμε εγκρίνει πολύ περισσότερες ουσίες, ιδίως νέες ενεργές ουσίες, λιγότερο επικίνδυνες, με χαμηλότερο δηλαδή προφίλ κινδύνου και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να εξασφαλίσουμε ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν να χορηγούν τις απαραίτητες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ιδίω για τις νέες χαμηλού κινδύνου ενεργές ουσίες. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην σωστή πορεία. Πρέπει ωστόσο να γίνει περισσότερη δουλειά στον συντονισμό και στην εναρμονίση των δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως και μεταξύ των χωρών μελών. Έχω και να θέσω ένα άλλο θέμα. Μιλήσατε για έκτακτες ή επίγουσες εγκρίσεις, το γεγονό ότι Πολλές από τις χώρες μέλη καταλήγουν σε αυτές διότι δεν έχουν αρκετέ ενεργέ ουσίε για να καταπολεμήσουν του επιβλαβεί οργανισμού. Αφενό αυτό είναι αληθέ, αλλά εν μέρη μόνο. Οι περισσότερε από τι επίγουσες εγκρίσει δίνονται για ουσίε οι οποίοι ήδη είναι εγκεκριμένε. Όχι επειδή δεν υπάρχουν μέσα προστασία των φυτών, αλλά απλώ διότι οι χώρε μέλη δεν έχουν πόρου για να δώσουν στις συνήθεις εγκρίσεις, των οποίων πρέπει να προηγηθεί μια σε βάθος αξιολόγηση. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ χωρών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον σκοπό αυτό εργάζεται, γιατί αυτό θα αποτελέσει και έναν από τους σημαντικούς πυλώνες του νέου κανονισμού προστασία των φυτών που ε, εκπονείται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από το 2009. Εν τέλει δε θέλω να θυμίσω την ε, ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα όπου θα εγκρίνονται διεθνώς οι ε, ουσίες. Και θέλω να σας επενθυμίσω ότι υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένα όρια περιεκτικότητας για να εξασφαλίζεται η ανοχή και είναι ο και υπάρχει ο κώδικας, ο σχετικός κώδικας, τον οποίον δέχονται οι χώρες μέλη. Βέβαια, η δυσκολία είναι ότι η έγκριση μιας ενεργού ουσίας δεν έχει σχέση μοναχά με την προστασία της υγείας του καταναλωτού, αλλά και με όλες τις ε, πτυχές της ε, υγείας, της έκθεσης δηλαδή στις ουσίες, της προστασίας του περιβάλλοντος και είναι πολύ δύσκολο να επιβληθούν τα πολύ υψηλά μας επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας σε τρίτες χώρες. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν τελειώνοντας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εγκρίνει τον κώδικα MRLs και επίσης ότι εργαζόμεθα προς την κατεύθυνση ενός, ε, της δημιουργίας ενός συστήματος συντονισμού για τις ελάσσονες χρήσεις για να λάβουμε υπόψη και την διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Θέλετε να λάβετε και εσείς το λόγο τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το άλλο θέμα που είχε τεθεί ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης νέων ασθενειών για τα φρούτα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά υπάρχουν στην Αφρική και 36 ε, κρούσματα σημειώθηκαν φέτος. Είναι γνωστό πρόβλημα. Συνεννοούμαστε εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια με την Νότια Αφρική για να γίνει κάτι. Δεν είναι πρώτη φορά όπως υπόθηκε και στο παρελθόν έγινε κάτι ανάλογο για την Αργεντινή και τη Βραζιλία και πάλι χρειάστηκε κάποιος χρόνος αλλά μετά από τα μέτρα άρχισαν να σέβονται και αυτοί τα κριτήρια μας για τις εισαγωγές. Πριν από ένα χρόνο αποφασίσαμε ότι αν υπάρξουν πάνω από πέντε κρούσματα και δεν ληφθούν μέτρα, τότε θα ληφθούν αντίμετρα από την Ένωση. Τέλη Αυγούστου σημειώθηκαν πέντε κρούσματα και γι' αυτό συνοηθήκαμε και στις αρχές Σεπτεμβρίου τους είπαμε χρειάζονται μέτρα. Που ήμασταν έτοιμοι και να τα προτείνουμε να τα εφαρμόσουν από την πλευρά τους. Μας το δέχτηκαν γραπτός, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα κρούσματα έγιναν γνωστά μετά και μας είπαν ναι αλλά τα φρούτα αυτά ε, δεν είχαν τύχει ακόμη των μέτρων αυτών. είχαν ήδη φύγει με τα πλοία πριν ληφθούν τα μέτρα. Ε, δεν μπορέσαμε να τα ελέγξουμε ακόμη όλα αυτά ακριβώς, αλλά τους είπαμε ότι υπάρχει αναφορά από την ομάδα εργασίας Γεωργίας και την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε μέτρα για την, ε, τον περιορισμό των εισαγωγών εσπεριδοειδών από την Νότια Αφρική μόνο και θα τις δεχόμαστε μόνο από περιφέρειες που είναι γνωστό ότι δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα. Αυτό έγινε δεκτό με μεγάλη πλειοψηφία και θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Όσο για του χρόνου, γιατί τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο την τωρινή περίοδο, δεν θα εφαρμόζονται για του χρόνου. Ζητήσαμε όμως από την ΕΦΣΑ να μας δώσει νέα επιστημονικά στοιχεία. Το έγγραφο που είδατε είναι, δεν είναι ακόμη τελικό. Το τελικό κείμενο θα το έχουμε τον Ιανουάριο και τότε θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν του χρόνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος Νομίζω ότι για τις συγκεκριμένες αναφορές νομίζω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, την οποία ακούσαμε τώρα, μας έδωσε ορισμένες εξηγήσεις σε σχέση με την καθυστέρηση της λήψης μέτρων γύρω από τις φυτοπροστατευτικές ουσίες οι οποίες προορίζονται για ελάσσονες χρήσεις ή για έκτακτες χρήσεις Αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο αφορά το σύνολο της ε, ε, φυτοπαραγωγής στην Ευρώπη. Έχοντας ακούσει πάντως τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να μάθω. Είναι σαν να μας λέτε ότι ναι μεν υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά και ότι σκοπεύετε να πάρετε κάποια μέτρα για την επόμενη εσοδεία, όχι για την παρούσα εσοδεία ιδιαίτερα με τα νοτιοαφρικανικά προϊόντα. Οι προβλέψει είναι μετριοπαθείς, θα ήθελα όμως να πω ότι η εμφάνιση της συγκεκριμένης αυτής ασθένειας θίγει τα προϊόντα από τη συγκεκριμένη χώρα και θα δημιουργήσει στην περίπτωση που επεκταθεί ε, πάρα πολλά προβλήματα γιατί πρόκειται για μια ασθένεια η οποία έχει τρομακτικές συνέπειες. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προλαμβάνει και να διασφαλίσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς από τη συγκεκριμένη αυτή ασθένεια. Τώρα η ΣΑΧΑ, η οργάνωση των παραγωγών, ζητά πιο συγκεκριμένα μέτρα άμεσα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια δίκαιη διεκδίκηση υποστηρίζεται από το κόμμα μου, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Απαιτείται μια απόλυτη και πλήρης αμοιβαιότητα σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες προϊόντων με ουσίες οι οποίες απαγορεύονται ε, στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον βέβαια έχουν τεκμηριωθεί οι ανάγκες για την έκτακτη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις ανάμεσα στο τι απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παραγωγή των άλλων χωρών, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συστηματικά οδηγεί στην απώλεια ανταγωνιστικής ικανότητας από πλευράς των Ευρωπαίων παραγωγών. Θα ήθελα λοιπόν ε, τα μέτρα αυτά να είναι μια μόνιμη ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια συστηματική ενασχόλησή της και για τους λόγους τους οποίους ήδη προανέφερα. Δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα, το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό η Ένωση Παραγωγών της Βαλένσια είχε ήδη παρουσιάσει μια πρώτη αναφορά το 2010 και το 2013 έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το ίδιο θέμα, την έλλειψη αντίδρασης δηλαδή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εκπροσώπους της μας είπε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός και τις επόμενες εβδομάδες θα ληφθούν μέτρα. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να δούμε ε, τι μέτρα ελήφθησαν ήδη από το 12 και μετά για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ασθένειες που έρχονται μέσα από την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση για μια ασθένεια η οποία δεν θα μολύνει μόνο ε, τα, την παραγωγή οποροφόρων αλλά θα δημιουργήσει και τεράστια προβλήματα πέραν αυτού υπάρχουν κάποια μέτρα ανοχής ανάλογα με το ποια είναι η χώρα. Είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και διαφορετική στάση ε, για κάθε χώρα. Πάντως το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση σε τέτοιου είδους καταστάσεις και θα πρέπει οι ισχυρισμοί ε, ε, της ε, Νοτιού Αφρικής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά με πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Υπάρχει ένα άμεσο πρόβλημα για την ασθενή αυτή μέσω των εξαγωγών και έχει ακριβώς τα στοιχεία που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει μέτρα. Η παραγωγή οποροφόρων ε, γενικά ε, στην, ε, στις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει λοιπόν μια ευθύνη φυσικά και συγκεκριμένα από τις χώρες που εξάγουν και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία μελέτη η οποία είχε ε, συγγραφεί ε, μέχρι το 2010 με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να μην μάλλον πάρουμε μέτρα και να απογοητεύσουμε τους γεωργούς και στην Ισπανία και στις άλλες χώρες. Ε... Κύριε Μπουστινάρου, αν είστε πολύ σύντομος παρακαλώ. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχαμε δύο τόσο συνδεδεμένες αναφορές τη Δροσόφυλα, Μελανογκάστερ και την Τωρινή. Κοιτάξτε πόσο γελοί γινόμαστε και λυπάμαι που το λέω. Φοβόμαστε την δροσόφυλλα και έτσι θέτουμε φραγμούς στην έρευνα αλλά δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο σημαντικό όπως την παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαστε με ένα θέμα που έχει τρομερές υγειονομικές συνέπειες και πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί ένα σύστημα επίγουσας ανάγκης όπου αν χρειάζεται να σταματάνε οι εισαγωγές ή να λαμβάνονται υγειονομικά μέτρα. Αν δεν υπάρχει κανένα σύστημα ταχείας αντιμετώπισης, τρία χρόνια αρκούν για την καταστροφή χιλιάδων εκταρίων γης ή και όλης της παραγωγής Ακόμη δεν ξέρουμε τις ακριβείς επιπτώσεις επί της υγείας. Έχουμε ναι. τόσα μέτρα και εργαλεία και τίποτα που να αφορά τόσο άμεσα ένα σοβαρό θέμα όπως της δημόσιας υγείας. Από την παρέμβαση του κ. Μποστινάρου το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίω είδαμε μια μεγάλη ευαισθησία και γνώση από τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Προτείνω να έχουμε ε, να ε, τεθεί στη διάθεσή μας ένα σύντομο κείμενο που να επεξηγεί στους αναφέροντες όλες τις δυνατότητες που, που τους παρέχει και όλες τις προοπτικές για την αναδιαμόρφωση της νομοθεσίας στα συγκεκριμένα θέματα ούτω ώστε να προστατέψουμε κάτι που είναι πιο σημαντικό ακόμη και από τη μίγα για την οποία μίλησε πριν ο κύριος ε, Μποστινάρου. Περιμένουμε λοιπόν πολύ σύντομα από την Επιτροπή μια παρουσίαση τελική, σύντομη, προκειμένου να την αξιοποιήσουν οι αναφέροντες και άλλοι που πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με τα ίδια ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη αναφορά του κυρίου Μάικλ Ρόλφ, Βρετανικής Ιταγένειας και τεσσάρων που τη συνυπογράφουν, σχετικά με την... Oh, sorry, yes. Señora Presidenta, muchas gracias, pero quiero que sepa que... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ένας διατροφικός κώδικς γενικά που προβλέπει όμως για τη χρήση ορισμένων ουσιών για αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων που όμως τις απαγορεύει οι Ηνωμένε Πολιτείες. Είμαστε πολύ αυστηροί για τη δροσόφυλλα μελανογκάστερ ενώ ταυτόχρονα πολύ χαλαροί για θέματα που απαιτούν καραντίνα ας πούμε και που αφορούν εκατομμύρια τόνους. Εδώ παίζουμε με τη φωτιά. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί, αλλά δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και έτσι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε μόνο μέσω των ε, έκτακτων αδειοδοτήσεων. Ζητάμε, απαιτούμε λύσεις τώρα που μας υποσχέθηκε και εμείς είμαστε μαζί σας να πιέσουμε όσο είναι δυνατό. Ε, λοιπόν, πάμε στην υπόθεση, στην καταγγελία του κ. Μάικλ Ρόλφ για ε, ασυμβίβαστα με βάση τη διατάξη του καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Κυπριακή νομοθεσία. Είναι εδώ ο κ. Ρόλφ. Ναι, παρακαλώ κύριε Ρόλφ. Madam Chair and uh, Committee Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και οι πέντε αναφέροντες προετοίμασαν την παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα. Κατανοούμε ότι λάβατε ένα αντίτυπο της παρουσίασης αυτής και των ε, προσθήκων της των παραρτημάτων. Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, οι Κυπριακέ Αρχέ είναι υπεύθυνε για τη ασφάλιση του γεγονότο ότι τα κτίρια πρέπει να είναι σαφή και σταθερά. Υπό το άρθρο 3 του Κυπριακού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κυπριακού Συντάγματο, είναι υπεύθυνοι εάν συμβεί κάτι σχετικά με αυτά. Τον Ιανουάριο του 2005 το Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών είχε καθορίσει ότι τα, οι κατοικίε μας είχαν πρόβλημα 150 χιλιοστών κίνησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους του, της Περιφερειακής Διοίκησης Πάφου στην Λευκοσία στις 7 Ιανουαρίου 2005 και φάνηκε εκεί ότι ο, δεν είχε γίνει τίποτα για να διορθωθούν τα πράγματα. Είπαν ρητά ότι είχαν αναλάβει την διόρθωση της κλίσης των κατοικιών μας. Είπαν ότι θα ήταν υπεύθυνοι και για την επιτήρηση της διόρθωσης και όρισαν τον κύριο Αγαπίου ως τον άνθρωπο που θα ήταν υπόλογος για όλα αυτά. Και τι έγινε μετά αντικαταστάθηκε ένας τείχος που χώριζε δύο σπίτια αλλά τίποτε άλλο για να διασφαλιστεί ότι θα σταθεροποιούνταν οι κατοικίες. Φαίνεται ότι ο κατασκευαστής είχε εκείνος καθορίσει τι θα έκανε και τι δεν θα έκανε ακολουθώντας και ο κύριος Αγαπίου απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες του. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί όπως ρωτήσαμε και εμείς. Και φάνηκε ότι ο κύριος Αγαπίου είχε σχέσεις συγγενικές με τον κατασκευαστή. Αφού μετά το 2005 ο κατασκευαστής έφυγε χωρίς να σταθεροποιήσει τις κατοικίες, ο κύριος Αγαπίου δεν ήταν πια σε θέση να μας πει τίποτα. Κατά τις επόμενες έρευνες μας μας είπαν ότι η διαφθορά είχε αναγκάσει όλους τους υπεύθυνους να παρατήσουν κάθε προσπάθεια. Όλα αυτά βέβαια ανησύχησαν ιδιαίτερα τους αναφέροντες, των οποίων οι κατοικίες τώρα έχουν κλείσει 190 χιλιοστά από μπρος προς τα πίσω. Είμαστε όλοι στη σύνταξη και καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερό πρόβλημα για μας η κλίση των κατοικιών μας που γίνονται σιγά σιγά άχρηστες τελείως. Και δαπανίσαμε χιλιάδες ώρες στις προσπάθειές μας. Οι αναφέροντες κυρίες και κυρία Μπρουκ είναι πάνω από 70 και δεν έχουν άλλο σπίτι εκτός από αυτό το οποίο κλείνει. Έχει καταστραφεί και η υγεία και η ευτυχία των. Αναγκαστήκαμε αυτόν τον εφιάλτη να τον υποστούμε πάρα πολύ καιρό και χρειαζόμαστε δική σας βοήθεια για να βρεθεί μια λύση για να μπορέσουμε να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας ήσυχοι. Καταλήγω και συνοψίζω. Το 2005 μας δόθηκε υπόσχεση ότι θα διορθωθούν οι κατοικίες μας, δεν έγινε τίποτα τέτοιο και υποστήκαμε πολλές ζημίες αλλά και στρες. Θέλουμε τη σταθεροποίηση των θεμελίων σύμφωνα με τα πρότυπα που λέει και η άδεια οικοδόμησης τη διόρθωση της κλίσης και όλα αυτά τα αναφέρει στην έκθεση του 2008 το ΙΤΕΚ. E e και όποτε δεν μπορεί να υπάρξει διόρθωση ζητούμε αποζημίωση. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε στη βοήθεια και στήριξή σας για να βρεθεί μια άμεση λύση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην ε, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον καταγγέλλοντα. Ε, προσπαθήσατε να, να βρείτε το δίκιο σας στον... Did you try to find your, you know, to compensate or to find your right by uh, appealing either to the uh, Cypriot uh, ombudsman Πρέπει να απευθύνεται έκκληση ίσως προς τον Κύπριο διαμεσολαβητή. Ή γενικότερα στην Κυπριακή δικαιοσύνη. Ναι, έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε πάει δύο φορές στον Κύπριο διαμεσολαβητή μας είπε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ τεχνικό για την υπηρεσία της και δεν μπορεί να ασχοληθεί. Και τι γίνεται με τα δικαστήρια. Δεν έχουμε πάει στα δικαστήρια. Γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει να καταγγείλουμε την Κυπριακή κυβέρνηση και να την παραπέμψουμε στα δικαστήρια. Όχι, εγώ ε, ίσως θα πρέπει να παραπέμψετε αυτούς οι οποίοι είναι οι κατασκευαστές μας είπαν ότι υπεύθυνοι υπεύθυνη για την αποκατάσταση είναι η Κυπριακή Κυβέρνηση από το 2005, οπότε αν προσφύγουμε θα πρέπει να προσφύγουμε εις βάρος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα στη θέση σας θα προσέφευγα στα δικαστήρια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εκφράζουμε τη λύπη και την συμπαράστασή μας προς τους αναφέροντες αλλά όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση μας τον Μάρτιο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Κομισιόν για αυτά. Το πρόβλημα της αναφοράς αυτής είναι θέμα εφαρμογής της νομοθεσίας για τον τομέα των κατασκευών και των οικοδομών που πρέπει να διασφαλίζει ότι θα εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες. Αφού τελειώσει η κατασκευή θεωρούνται έτοιμα τα κτίρια και δεν γίνεται πια τίποτα. Στην αρχική αναφορά σας μιλούσατε για ένα κυπριακό νομοθέτημα του 2009. Η οδηγία που αφορά τα κτίρια από το, από το περιεχόμενο της αναφοράς σας φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται εδώ, αλλά Πρέπει ο κατασκευαστής και η κυπριακή κυβέρνηση να αποκαταστήσουν τις ζημίες, αν υπάρχει ζημία στα θεμέλια. Εκτός αυτού, η οδηγία για τις παράνομες εμπορικές δραστηριότητες ή πρακτικές διαφέρει, δεν είναι το ίδιο πράγμα γιατί αφορά θέματα ασφαλείας των πολιτών. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν βλέπεις και κανένα λόγο να συνεχίσει την περίπτωση αυτή και σας ε, προσκαλεί να έρθετε σε επαφή με κυπριακές οργανώσεις για να πάρετε νομικές συμβουλές. Είναι και οικονομικό όμως το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Βάτσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο κυρία Πρόεδρε γιατί ο κύριος Ρόλφ προέρχεται από την εκλογική μου περιφέρεια και έχω παρακολουθήσει με ενδιαφέρον εδώ και μερικά χρόνια την υπόθεσή του και το παράπονο του καθώς και της οικογένειας Μπρούξ και Ράντφορντ. Υπάρχει παρόν εκπρόσωπος της Κυπριακής Μόνιμης Αντιπροσωπείας σήμερα. Βρίσκω ότι πρόκειται για έσχος οι μόνιμες αντιπροσωπείες γνωρίζουν καλά τις σημερινές διατάξεις, των επιτροπών μας και με τέτοιο θέμα θα έπρεπε σίγουρα να είχαν στείλει εκπρόσωπο. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε στο μέλλον να τους ζητήσετε να στείλουν εκπρόσωπο όταν εμφανίζονται στις ημερήσεις διατάξεις τέτοια θέματα. Οι ψηφοφόροι μου έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες μετά την ε, αγορά των κατοικιών τους. Ολόκληρη λίστα ζημιών ένας τείχος που υποτίθεται ότι θα εμποδίσει τις κατοικίες να αρχίσουν να τσουλάνε προς τα κάτω, κατέρευσε το 2004 που είχε χτιστεί πρώτα χωρίς άδεια και μόνο με μεγάλη πολιτική πίεση κατάφεραν να αναγκάσουν τους κατασκευαστές να ε, ξαναανεγείρουν τον τείχο αυτό. Και μετά ανεκάλυψαν ότι ο σχεδιασμός των κατοικιών δεν συμμορφωνόταν με την ε, άδεια ε, οικοδόμησης αλλά ήταν σε πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές. Και εκεί θα έπρεπε να είχε δράσει η ε, κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτησίες αυτές είναι αδύνατο να απολυθούν διότι είναι ανασφαλείς. Γνωρίζω ότι το άρθρο 345 της συνθήκης αποκλείει θέματα εγγύου ιδιοκτησίας από τις αρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό και βασίζονται στις διατάξεις περί αθέμητου ανταγωνισμού. Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν σαφή, Άλλωστε, δόθηκε υπόσχεση από το Υπουργείο Ιστορικών, όπω ακούσαμε και από τον ίδιο τον Ρόλφ, από το Υπουργείο Ιστορικών, λέγω, της Κυπριακή Δημοκρατίας, που δεν ε, την σεβάστηκε τελικά. Και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενιαία αγορά. Και η ενιαία αγορά προσφέρει στους πολίτε την ελευθερία να αγοράσουν κατοικία όπου επιθυμούν και να εγκατασταθούν όπου επιθυμούν. Εάν όμω η νέα αγορά δεν του προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους προσφέρει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παρόμοια με αυτήν που θα μπορούσαν να μένουν στις ίδιες τις χώρες μέλη τους, τότε η Ένωση εγκαταλείπει τους πολίτες. Η ενιαγορά αγορά προϋποθέτει ότι οι αγορές που έγιναν κάπου αλλού θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη εφόσον υπάρξουν προβλήματα. Γι' αυτό θα ήθελα ο αρμόδιος επίτροπος να θέσει το θέμα υπόψη της Κυπριακής Κυβερνήσεως. Αν δεν το έχει πράξει ο αρμόδιος επίτροπος, θα το πράξει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας αυτού. χωρίς οι ίδιοι να χρειαστεί να αναλάβουν δαπανηρές και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Γι' αυτό και υποβάλλω αίτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ εσά η Κομισιόν να ζητήσει από το ύψιστο δυνατό επίπεδο να παρέμβουν στην Κυπριακή Δημοκρατία για να ζητήσουν δικαιοσύνη για τους αναφέροντες. I completely agree with you, uh, dear colleague, and I can understand. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι προφανές ότι οι κάτοικοι των σπιτιών αυτών υφίστανται μεγάλο στρες, αλλά πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν απευθύνθηκαν στην Κυπριακή δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για να διαφωνήσω σαφιστούν τα πράγματα. Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία έμαθε για το θέμα. Δεν μπορούσαν να έρθουν, δεν θέλαν να έρθουν σήμερα, δεν ξέρω, αλλά αποφασίσαμε εδώ να στείλουμε μία επιστολή σε επίτροπο και στον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου για να πάρουν κάποια θέση επί του προβλήματος. Μήπως η Κομισιόν μπορεί να βρει και κάποια εναλλακτική α, και άλλη μια λύση. Αν βρείτε τρόπο να πιέσουμε την Κυπριακή κυβέρνηση θα ήταν θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτε άλλο. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Απλώς ευχαριστούμε. Δεν έχουμε τώρα τίποτα. Α, έχουμε, έχουμε. Του κυρίου Βαλέσα, που δεν έχει πολύ χρόνο, αλλά έχει. Ναι. Επειδή έχουμε μόνο πέντε λεπτά, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Και μόνο δύο συναδέλφους. Οπότε θα τα πούμε άμεσα. Τρία πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε. Πρώτον, είναι η τελευταία ετήσια έκθεση της Επιτροπής μας σε αυτή τη θητεία και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να περιγράφει και τις δραστηριότητε της Επιτροπής μας το 2013 αλλά να κάνει και μια γενικότερη περιγραφή της θητείας. Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς καταφέραμε και κατά πόσον να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών, ιδιαίτερα με τις νέες δικαιοδοσίες που μας δίνει η καινούργια συνθήκη. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε νέες συστάσεις ως προς το πώς θα μπορούσε η εργασία της Επιτροπής μας να γίνει πιο αποτελεσματική, όχι μόνο εδώ μέσα, αλλά και σε συνεργασία με άλλα όργανα όπως την Κομισιόν, και τον διαμεσολαβητή. Και θα έπρεπε επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τις εθνικές αρχές. Αυτή είναι η γενική μου περιγραφή. Όσο για τη δομή του εγγράφου αυτού της έκθεσης, πρέπει νομίζω να έχει τρία ή τέσσερα μέρη. Πρώτον, τις δραστηριότητες του τελευταίου έτους του 2013. Και μετά ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς μας. Να δούμε τι ακροάσεις γίνανε, τι ειδικέ ε, εκθέσεις στην εκλογή του διαμεσολαβητή και επίσης των συστάσεων των προηγούμενων ετήσεων εκθέσεων. Και μετά να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και στην αναγκαιότητα αναθεώρησης των, του εσωτερικού μας κανονισμού. Να το αναλύσουμε αυτό ιδιαίτερα. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τη συνεργασία μας με το διαμεσολαβητή. Μέσω μιας νέας διαθεσμικής συμφωνίας να δούμε πώς θα μπορούμε να ασχοληθούμε και με τα εθνικά δίκτυα των διαμεσολαβητών αυτά. Αυτά. Ορίστε κύριε Ποστινάρο, επειδή είμαστε μόνον τρεις, θα ήθελα να σας πω ότι δέχομαι την περιγραφή και το περιεχόμενο αυτό. Δεν θέλω όμως να ξεχαστεί η ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ξέρω ότι μόλις τώρα άρχισε να εφαρμόζεται και θα μας δοθεί ως θα τη δώσουμε ως κληρονομιά στους επόμενους βουλευτές. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι βάση για μελλοντική τους έμπνευση. Να προσθέσω κάτι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, αν και δεν είναι δικιά μου η ιδέα, αλλά της κυρίας Ρέιλι όταν ε, ήρθε εδώ να είχε πει ότι υπάρχει Επιτροπή Αναφορών και στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ίσως ο καθένας από μας θα έπρεπε να ζητήσει ανάλογες επιτροπές αναφορών να καθοριστούν σε όλες τις βουλές των κρατών μελών. Αυτή την ιδέα ήδη την εξέφρασα και στο, στη δική μας Βουλή, στη δική μου, αλλά εμείς όλοι ως μέλη της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να το διαδώσουμε αυτό ως ιδέα στους εθνικούς βουλευτάς, διότι είναι δουλειά πολύ πιο σοβαρή από ό,τι των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. κοιτάξτε, χαίρομαι ιδιαίτερα η πρόταση αυτή συμφωνεί και με τις δικές μου σκέψεις ως προς την πρωτοβουλία των βουλευτών. Θα τη βάλω, φυσικά θα τη βάλω. Ωραία. Τώρα. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία προτείνεται να αφαιρεθούν από τις αναφορές που θα κλείσουν. 15 και 16 του καταλόγου που έχετε. Η μία προέρχεται από την Ισπανία και αφορά τις χωματερές κοντά σε πόλεις. Και άλλη μία επίσης από την Ισπανία που αναφέρεται στις 22 Ιουλίου σαν Ευρωπαϊκή ημέρα για τα μνήμης για τα θύματα του μίσους. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μειοψηφία είμαστε, λέει η πρόεδρος. Have a nice weekend. I close the meeting. <laughs> Ε,